Καλησπέρα. Αντικαθιστώ τον συνάδελφο Μπούζεκ. Είδατε το πρωί ότι δεν αισθανόταν πολύ καλά και λόγω της ε, αρρώστιας του ε, επιστρέφει στην πατρίδα του. Πρώτο θέμα είναι πρόταση οδηγίας του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας που αφορούν τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου. Ο κύριος Μπούζεκ επρόκειτο να, παρουσιάσει το θέμα αυτό. Ωστόσο, μιας και δεν είναι εδώ, θα τον, ε, θα τον αντικαταστήσει ο κύριος Κάριντς. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφοι. Μιλώ εκ μέρους του Ζέρζι Μπούζικ. Γι' αυτό και θα διαβάσω τα σημειώσει που εκείνος είχε προετοιμάσει. Χαιρετίζουμε την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της πρότασης για την τροποποίηση της οδηγίας για το φυσικό αέριο του 2009. Εγώ επίσης χαίρομαι που ο κύριος Κλάους Ντίτερ Μπόλχαρντ, ο διευθυντή ε, τη ε, Κομισιόν είναι εδώ μαζί μας και νομίζω ότι θα είναι σε θέση να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματά σας. Η πρόταση αυτή έχει τεχνικό χαρακτήρα και περιορισμένο εύρος. Και παρότι ε, ορισμένοι ισχυρίζονται ότι η ισχύουσα νομοθεσία ρυθμίζει ήδη τα ζητήματα αυτό, η νομοθεσία αυτή, οι διατάξει τη είναι ασαφή και πολλέ φορέ υπάρχουν παρερμηνίε. Γι' αυτό και στο Κοινοβούλιο πολλέ φορέ έχουμε καλέσει την Κομισιόν να συμπληρώσει και να καλύψει αυτό το νομοθετικό κενό. Και χαίρομαι που αυτό πλέον γίνεται. Σημειώνουμε ότι οι κανόνε Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, συμπεριλαμβανομένης της αποδέσμευσης, της ε, πρόσβασης τρίτων και της διαφάνειας θα πρέπει να ισχύουν για όλους τους αγωγούς από και προς τρίτες χώρες έως και ε, την, έως τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι σημαντικό για να εξασφαλιστεί ο θεμετός ανταγωνισμός ε, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η ασφάλεια των προμηθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ασφάλεια λοιπόν και η διαφάνεια στον τομέα του φυσικού αερίου θα παρέχουν βεβαιότητα και σαφήνεια καθώς και προβλεψιμότητα. νομίζω ότι αυτά είναι βασικά στοιχεία για κάθε ειλικρινή ε, επενδυτή ή φορέα που θέλει να ε, τηρεί δίκαιους, τους δίκαιους κανόνες. Τα στοιχεία αυτά ωστόσο είναι ζωτική σημασία και για τον κλάδο αλλά και για τους πολίτες. Ενισχύουν τον ανταγωνισμό και καταλήγουν σε χαμηλότερες τιμές χωρίς διακρίσεις για όλους τους καταναλωτές. Και τέλος είναι σημαντικό για τον ανταγωνισμό και την ανθεκτικότητα για, για την ολοκλήρωση μάλλον και την ανταγωνιστικότητα της ενεργειακής μας ένωσης βάσει αρχών και αξιών και όχι εξαιρέσεων. Η ετήσια έκθεση σχετικά με την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης θα παρουσιαστεί στην μικρή σύνοδο Ολομέλειας που θα γίνει αύριο, που θα επικεντρώσει στις διασυνδέσεις μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις ε, αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, πρέπει να μας απασχολήσουν και ζητήματα προμήθειας φυσικών αερίων από τρίτες χώρες, κάτι που καθώς οι εισαγωγές ανέρχονται σε περίπου 70% στην Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικού αερίου. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να δοθεί ορισμός στον φορέα διασύνδεσης ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών. Με την πρότασή της η Κομισιόν λοιπόν ε, βοηθά στο να εξασφαλιστεί η συμβατότητα των ε, αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Προφανώς, όπως και με κάθε νομοθέτημα, ανακύπτουν ορισμένα ερωτήματα. Πρώτον, ανάγκη να εφαρμοστούν νέοι κανόνες σε όλους τους νέους αγωγούς. Έχω ακούσει ότι από κάποιους, κάποιες αντιρρήσεις, ενώ ακούγεται ότι ε, ενδέχεται να τεθεί σε κίνδυνο το δικαίωμα των κρατών μελών να χορηγούν εξαιρέσεις. Δεύτερον, σε ποιο βαθμό ε, η πρόταση της Κομισιόν εξασφαλίζει όλους τους στόχους της ε, Ενεργειακής Ένωσης. Εγώ ως συζητητής Είμαι ανοιχτός σε όλα τα ερωτήματα και θέλω να ε, συζητήσουμε όλες τις ε, αμφιβολίες που έχουν εκφραστεί. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι η πρόταση Κομισιόν ανταποκρίνεται στις γενικές μας απαιτήσεις και εξυπηρετεί τους στόχους που έχουμε θέσει. Ευχαριστώ για τους σοσιαλιστές, ο κύριος Νίκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να χαιρετήσω τα όσα είπε ο συνάδελφος, ο κύριος Μπούζεκ, μέσω του εκπροσώπου του βέβαια εδώ πέρα, και θα ήθελα να εκφράσω και τη δική μου την άποψη. Το ότι, το, το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να τροποποιήσει την ε, οδηγία αυτή προκειμένου οι κανόνες που έχουν να κάνουν με τη μεταφορά φυσικού αερίου μεταξύ ενός ή και περισσότερων κράτων μελών θα έχουν να κάνουν πλέον και με τις τρίτες χώρες, είναι κάτι το ιδιαίτερα θετικό και χαίρομαι πραγματικά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία. Πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε ότι πραγματικά χρειαζόμαστε μια εσωτερική αγορά ενέργειας, στα πλαίσια της οποίας η ενεργειακή ασφάλεια, η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού θα είναι στοιχεία κεντρικά, κεντρική σημασία. Χρειάζεται λοιπόν ασφάλεια εφοδιασμού και διαφοροποίηση βέβαια των ενεργειακών πηγών, γιατί σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να ζήσουμε εδώ πέρα στην Ευρώπη την εμπειρία που είχαμε πριν από μερικού χειμώνε. Θα θυμάστε την εποχή εκείνη δηλαδή που τον έχει κανείς θέρμανση ακόμα και στο σπίτι του ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο και επισφαλές για πάρα πολλούς Ευρωπαίους πολίτες. Χρειαζόμαστε μια ανταγωνιστική αγορά, μια αγορά που να λειτουργεί καλά στην πράξη και που να προσφέρει δίκαιες τιμές για όλους τους καταναλωτές και που να συνάδει ουσιαστικά με την υφιστάμενη νομοθεσία. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι ε, η πρωτοβουλία αυτή της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ουσιαστικά ενισχύει περισσότερο την αρχή της ενεργειακής αλληλεγγύης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αρχή, η οποία όπως ξέρετε είναι πάρα πολύ σημαντική και ουσιαστικά έρχεται να ανταποκριθεί σε πάρα πολλές εκκλήσεις που έχουν κάνει τα κράτη-μέλη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρετε, το ζήτημα αυτό μας έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Η ενεργειακή ασφάλεια πρέπει και είναι ένα κοινό αγαθό. Χαιρετίζω λοιπόν την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συμφωνώ με το φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα που μας παρουσιάστηκε και ελπίζω να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό. Σας ευχαριστούμε κύριε Νίκα που σεβαστήκατε το χρόνο αγόρευσης. Ο κύριος Κναστοντεύσκη τώρα για το ECR παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αποφασιστικότητα την οποία έδειξε υποβάλλοντας την πρωτοβουλία αυτή και θέλοντας τελικά να ξεκαθαρίσει το νομικό καθεστώς που διέπει τους αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου. Όπως ξέρετε και ενδεχομένω θα πρέπει να στο επενθυμίσω ποιο είναι το πολιτικό πλαίσιο του ολοζητήματος. Αναφερόμαστε εδώ πέρα σε κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη συμβολική σημασία. Το ζήτημα είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και ιδίως βέβαια για όλους εκείνους που κατοικούν στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Και σε ελπίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα υποκύψει στην πίεση που ασκούν τα λεγόμενα ισχυρά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται αυτή τη στιγμή ιδιαίτερα αποφασισμένη να υπερασπιστεί τι μικρέ και πιο αδύναμε χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζουμε και ότι προκειμένου θα δείξει την ίδια αποφασιστικότητα υπερασπιζόμενη τις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές στην περίπτωση στον τομέα της Ενεργειακής Ένωσης αυτή τη φορά. Ξέρουμε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στα πλαίσια του Συμβουλίου. Δυστυχώς το Συμβούλιο δεν έχει δώσει ακόμα συγκεκριμένη εντολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια μικρή μειονότητα η οποία μπλοκάρει την όλη διαδικασία και επιβραδύνει το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εδώ στην Επιτροπή ΙΤΡΕ θα κάνουμε πάντως κάθε το δυνατό προκειμένου να ολοκληρώσουμε την εργασία που στην αναλογεί το συντομότερο δυνατό. Κάτι ακόμα. Ακούμε δεξιά και αριστερά κάποια επιχειρήματα από τη Γερμανία για παράδειγμα και από κάποια άλλα κράτη-μέλη τα οποία λένε ότι είναι έτοιμα να στηρίξουν τις προτάσεις αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αναφέρονται εδώ πέρα στην δυνατότητα να μπορεί κανείς να επιλέγει το ενεργειακό του μείγμα για λόγους ενεργειακής ασφάλειας. Αναφερόμενο εδώ πέρα και στάση από κύριο Κάριν, θα ήθελα να πω ότι ιδίω όσον αφορά τον τομέα τη ηλεκτρική ενέργεια υπάρχουν και συγκεκριμένοι στόχοι όχι μόνο ενεργειακή και ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και στόχοι καταπολέμηση ή μετριασμού μάλλον των κλιματικών αλλαγών. Επομένω, το ζήτημα δεν έχει να κάνει μόνο με μεταφορά από μια τρίτη ουδέτερη χώρα, Ουσιαστικά αναφερόμαστε εδώ πέρα σε μεταφορά φυσικού αερίου από μια χώρα επί της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει κυρώσεις και η οποία έχει προκαλέσει σύγκρουση και πόλεμο στην άμεση ανατολική γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ε, τα όσα λέγονται εδώ πέρα και απευθύνομαι προσωπικά και στον Πρόεδρο, τα όσα ακούσαμε έρχονται σε άμεση αντίθεση με τις βασικές αρχές που υποτίθεται ότι δημοσίως προασπίζεται η χώρα από την οποία προέρχεστε. Πάντως, και αυτό αποτελεί συμβολικό παράδειγμα ότι όλα αυτά τα οποία λέγονται δεν αποτελούν πάντα πραγματικότητα. Κύριε Κρασνοστεύσκη, με αναφέρετε, εγώ συμφωνώ μαζί σας και όχι με την κυβέρνησή μου. Ο κύριος Πίτερσεν από την Άλτε, που καθιστεί τα κύριο Φίνελε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Λέω ο κύριος Πέτρεσαν, θα είμαι πολύ σύντομος. Νομίζω ότι η περιγραφή που ακούσαμε ήταν ήδη πολύ καλή. Βλέπουμε ποιο είναι το όλο υπόβαθρο της πρότασης και για ποιο λόγο τελικά είναι αναγκαία. Πέρα από την βελτίωση του εφοδιασμού σε φυσικό αέριο, Λέγεται εδώ πέρα και κάτι το οποίο είναι προφανές, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται πάρα πολύ από εισαγωγές φυσικού αερίου από τρίτες χώρες θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εκτενέστατη συζήτηση για το αν η εισαγωγή φυσικού αερίου είναι η καλύτερη μακροπρόθεσμη λύση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντω σίγουρα θα είναι μια λύση την οποία θα πρέπει να αποδεχτούμε και για τα επόμενα χρόνια, για πολλά χρόνια ακόμα στο μέλλον. Και ακριβώς όπως λέγεται εδώ πέρα στην πρόταση αυτή ότι το κοινοτικό δίκαιο ισχύει για την δικαιοδοσία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τα χωρικά ύδατα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προβλέπεται εφαρμογή στις παροχές από τρίτες χώρες. Ακριβώς λοιπόν αυτές τις τρίτες χώρες θέλουμε τώρα να καλύψουμε την πρόταση αυτή και να καταφέρουμε τελικά να έχουμε περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά και τι μεθόδους που χρησιμοποιούν αλλά και άλλε βασικές αρχές όπως η κατάρτιση των τιμών και το καθεξής. Όπως ακριβώς λοιπόν το κάνουμε σε άλλους κλάδους, έτσι και στον τομέα της ενέργειας θα πρέπει να έχουμε το, κάτι το ανάλογο. Κάθε φορά που συζητάμε τέτοια ζητήματα όπως τώρα αγωγή φυσικών αερίων από και προς τρίτες χώρες. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που διεξάγεται τώρα αυτή η συζήτηση και που μας απασχόλησε και τα προηγούμενα χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μετά από όλες αυτές τις συζητήσεις βλέπουμε επιτέλους μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πραγματικά ελπίζω ότι και στο Συμβούλιο θα γίνουν ανάλογες συζητήσεις για το ζήτημα αυτό. Τέλος, ε, όσον αφορά το Nord Stream 2, νομίζω ότι ε, ακούστηκαν κάποιες απόψεις ότι ε, και για μένα και για κάποιους άλλους και γενικότερα για τις επιτροπές θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις του αγωγού αυτού για τις τιμές φυσικού αερίου. Ακούγονται διάφορα σενάρια όσον αφορά την κατάρτιση των τιμών. Αυτή τη στιγμή ολοκληρωθεί το σχέδιο Nord Stream 2. Νομίζω το ζήτημα αυτό δεν το έχουμε θίξει αρκετά και Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε και αφού το καλύψουμε εκτενώς σε μελλοντικέ μας συζητήσει, προκειμένου να μπορούμε να αξιολογήσουμε μελλοντικά σενάρια κατάρτιση τιμών στον τομέα του φυσικού αερίου παντού στην Ευρώπη. πάντω οι εξελίξει από ό,τι φαίνεται είναι θετικές και όπω και οι υπόλοιπε πολιτικές ομάδες στηρίζουμε και εμεί αυτή την πρόταση. Ο κ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρόθεση μια τόσο σημαντική πρόταση όπω είναι η τροπήση τη οδηγία για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου. Το ελάχιστο που επιβάλλει είναι να δοθεί ο απαιτούμενο χρόνο για σοβαρή επεξεργασία του κειμένου και σωστή προετοιμασία. Η διαδικασία του κατεπήγοντο που έχει προταθεί πλήττει τόσο τη δουλειά που επιβάλλεται να γίνει, όσο και το κύριο τη Επιτροπή μα, που για ένα τόσο σοβαρό νομοθετικό κείμενο επέλεξε τη συνοπτική διαδικασία. Δυστυχώ, η ίδια προχειρότητα έχει επιδειχθεί και από την Κομισιόν. Είναι απαράδεκτο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει την πρότασή τη χωρί να εκπονήσει μελέτη εκτίμηση των επιπτώσεων. Α μην ξεχνάμε πω η Κομισιόν έχει δεσμευτεί να εκπονεί μελέτη εκτίμηση των επιπτώσεων για όλα τα νομοθετικά μέτρα που προτείνει. Ιδιαίτερα δε για αυτήν την νέα πρόταση, δεδομένων των σοβαρών επιπτώσεων που μπορεί να έχει, απαιτείται σαφή νομική ανάλυση και μελέτη εκτίμηση των επιπτώσεων ακόμη και εξέταση του ενδεχομένου σύγκρουση με το διεθνέ δίκαιο. Η ομάδα τη Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά δεν θα στηρίξει μια πρόταση που βασικό στόχο έχει να ακυρώσει τα κυριαρχικά δικαιώματα και τι εξουσίε των κρατών μελών σχετικά με του όρου εκμετάλλευση των ενεργειακών του σπόρων. Τα δικαιώματα αυτά των κρατών απορρέουν τόσο από την ίδια τη συνθήκη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από το διεθνέ δίκαιο. Δεν γίνεται να μην λαμβάνουν υπόψη οι ιδιαιτερότητε που υπάρχουν σε κάθε κράτο, οι οποίε και καθιστούν αναντικατάστατον τον ρόλο των επιμέρου εθνικών πολιτικών στην ενέργεια. Ιδιαίτερα να είναι ευέλικτε αυτέ οι, οι πολιτικέ. Η προσπάθεια χειραγώγηση των κρατών μελών σχετικά με την άπτυξη συναγωγών με τρίτε χώρε, το μόνο που θα επιτύχει είναι να οξυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ένωση όσον αφορά την ενεργειακή τροφοθεσία και ασφάλεια. Στα σοβαρά ενεργειακά προβλήματα και αδιόξοδα που ταλανίζουν του λαού, η Κομισιόν απέτυχε και πάλι να προτείνει ουσιαστικά μέτρα. Χαρακτηριστικό αποτελεί το γεγονό πω δεν έγινε καμία προσπάθεια να ενισχυθεί η πρόταση όσον αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών σε σχέση με το φυσικό αέριο. Ούτε κατατέθηκε μέχρι σήμερα ολοκληρωμένο σχέδιο για ανάπτυξη και αξιοποίηση των εχώριων πηγών φυσικού αερίου τη Ένωση, όπω είναι για παράδειγμα τα σημαντικά κοιτάσματα που ανεβρέθηκαν στην Ανατολική Μεσόγειο. Δυστυχώ, εκεί που δόθηκε όλη η σημασία, κατά την άποψή μα, ήταν να προωθηθούν με ταχύτητα οι απαιτούμενε αλλαγέ, ώστε να τεθεί φραγμό στο Nord Stream 2. Και εδώ είναι το λάθο που πιστεύουμε ότι κινείται η Επιτροπή και ενδεχομένω να κινηθεί και το ε, Κοινοβούλιο να εθετήσουμε ε, μια τέτοια οδηγία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Σιλικιώτη. Τέσσερις άλλους συναδέλφους θα ακούσουμε τώρα. Θα ήθελα να μιλήσουν για αυτό το θέμα. Για ένα λεπτό ο καθένας. Σας ενθαρρύνω παρακαλώ να σεβαστείτε το χρονοδιάγραμμα, γιατί είμαστε πολύ πιεσμένοι χρονικά. Η κυρία Βέρνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω μεγάλες αμφιβολίες όσον αφορά την ε, νομική βάση αυτής της πρότασης. Οι νομικές υπηρεσίες της Κομισιόν και του Συμβουλίου κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει νομική βάση για την αναθεώρηση της οδηγίας για το φυσικό αέριο. Και αυτό που με ανισχύει ακόμα περισσότερο είναι το γεγονό ότι δεν έγινε διαβούλευση από πλευρά Κομισιόν με του εμπλεκόμενου φορεί και του ενδιαφορεμένου, ούτε μελέτη επιπτώσεων. Και αυτό παρά το γεγονό ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ουσιώδη τροποποίηση τη οδηγία διότι απαιτούμε πλέον οι κανόνες εσωτερικής αγοράς να ισχύουν και σε τρίτες χώρες. Και αυτό είναι σημαντική αλλαγή που θα έχει σημαντικές επιπτώσεις και όσον αφορά τον εφοδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς το κανονιστικό πλαίσιο πλέον δεν θα αφορά μόνο το Nord Stream 2, αλλά και όλους τους πιθανούς μελλοντικούς αγωγούς. Επίσης, θα με ενδιέφερε ο κύριος, αυτό που είπε ο κύριος Φέντερ, λέει ο κύριος Πέτερσεν. Υπάρχει μελέτη αντικτύπου πώς τελικά έχουν επηρεαστεί οι τιμές του φυσικού αερίου. Κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό και ενδιαφέρον για τους πολίτες μας. Νομίζω ότι πρέπει να οδηγηθούμε σε μια ειλικρινή εκτίμηση της κατάστασης. Η Ρωσία μέχρι τούδε έχει αποδειχθεί ότι είναι ένας αξιόπιστος προμηθευτής και η εξάρτηση ε, έχει έναν διτό χαρακτήρα, έναν αμοιβαίο χαρακτήρα. Και εμείς θέλουμε το φυσικό αέριο της Ρωσίας, αλλά και η Ρωσία χρειάζεται τα ευρωπαϊκά χρήματα. Άρα, αν ε, τελικά διακοπεί η σύνδεση από την Ρωσία από πού θέλουμε να τροφοδοτούμαστε με φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν, από άλλες χώρες της ε, Ανατολικής Ευρώπης ή μήπως από ε, τις ΙΠΑ, ε, από, φρακ, ε, από ε, υδρορογμάτωση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς καλωσορίζω την πρόταση της Κομισιόν και συμφωνώ με τους στόχους της. Πρέπει να είναι σαφέστερος ο κανονισμός πρέπει να είναι πιο ακριβής και ο γενικός στόχος πρέπει να παραμείνει ο ίδιος. Η αύξηση της ε, ασφάλειας ανεφοδιασμού, ειδικά στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Μιλήσαμε για το πόσο δύσκολο είναι τις, τις ε, χειμωνιάτικες μέρες να μην έχουμε παροχή φυσικού αερίου. Μία ερώτηση για το πεδίο εφαρμογή της πρότασης. Καλύπτει τους αγωγούς που περνούν τα χερσαία σύνορα π.χ. μεταξύ Ουκρανίας και Ουγγαρίας. Γιατί δεν νομίζω ότι το κείμενο είναι αρκετά σαφές σε αυτό το επίπεδο. Και μια άλλη ερώτηση σε ό,τι αφορά τις τρίτες χώρες. Πρέπει να κάνει μια διαφοροποίηση ανάμεσα στις χώρες που ανήκουν στην ενεργειακή κοινότητα γιατί έχουν ευθυγραμμίσει τους κανονισμούς του με τους δικούς μας πολύ περισσότερο από ό,τι άλλες τρίτες χώρες. Προτείνω λοιπόν τα μέλη της ενεργειακής κοινότητας να τύχουν διαφορετική ε, μεταχείρισης. Ε, θα μιλήσω εξ ονοματό μου, λέει ο κύριο ε, Κάριτς. απόλυτη υποστήριξη της πρότασης της Κομισιόν. Ούτε 30 δευτερόλεπτα σας πήρα. κύριος Ευχαριστώ. Εν πάση περιπτώσει, ε, κυρώσεις, ενεργειακή κοινότητα, αλληλεγγύη, σε ποιο θέμα τελικά αναφέρεστε, δεν γνωρίζετε ποια είναι η πραγματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να έχει απόθεμα φυσικού αερίου ε, για τουλάχιστον 30 μέρες, τουλάχιστον. Και υπό ορισμένες συνθήκες η υποχρέωση αποθήκευσης ε, φυσικού αερίου είναι ακόμα μεγαλύτερες. Τι θέλετε, εν πάση περιπτώσει, να περιορίσετε την εθνική κυριαρχία των κρατών μελών. Γιατί δεν υπάρχουν αντίστοιχοι κανόνες για τις εισαγωγές πετρελαίου, ξυλία, λιγνίτη. Γιατί λοιπόν ε, δεν ε, ισχύουν τέτοιου είδους κανόνες για, όλους, ε, για όλες τις πηγές ενέργειας από άνθρακα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κακή η πρόταση. Έχει έναν και μόνο στόχο και αυτός είναι να εμποδίσει στην πραγματικότητα τα κράτη-μέλη να διαμορφώσουν και να χαράξουν τη δική τους ενεργειακή πολιτική. Ο διαχωρισμός, το unbundling, έχει αποδειχθεί περίτρανα ότι είναι πέρα για πέρα αναποτελεσματικός. Και ξαναλέω, γιατί δεν εισάγουμε τέτοιους κανόνες και για άλλα αγαθά, πετρέλαιο, λογνίτη κτλ. κτλ. Μήπως κάπως ε, έτσι καταφέρουμε να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο την ε, δημοφιλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. The... Κάνετε μερικές ερωτήσεις. Ο... Το άτομο από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας θα μπορούσε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα μπορούσε να σας απαντήσει ε, σε αυτές τις ερωτήσεις και στις ερωτήσεις των υπολείπων. Έχετε το λόγο, πρόσωπε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να ξεκινήσουμε με την τελευταία ερώτηση, γιατί με αυτή μπαίνουμε στο ψητό της ε, λογικής και του γιατί υποβάλαμε αυτή την πρόταση. Ο κύριε Κούλιτσε, δεν θέλουμε προφανώς να παρεμποδίσουμε τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν ενεργειακή αποδοτικότητα ή όπως άκουσα να λέγεται να παρέμβουμε στο ενεργειακό μείγμα και στην επιλογή του ενεργειακού μείγματος των κρατών μελών. Αυτή η πρόταση δεν πάει τόσο μακριά. Αυτό που κάνει, και το είπαν και πολλοί συναδελφοί σας πήραν το λόγο, είναι ότι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ασφάλεια δικαίου και σαφήνεια νομική για το νομικό καθεστώς που διέπουν τους αγωγούς και που ξεκινάνε από τρίτες χώρες και μπαίνουν ε, σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιο είναι το καθεστώς που τους διέπει. Αυτή η πρόταση δεν επιτρέπει στην Κομισιόν ή σε οποιοδήποτε άλλο θεσμικό όργανο να παρέμβει στο αν ή όχι θα χτιστεί ας πούμε, ένας, ένας αγωγός ε, φυσικού αερίου. Αυτό που κάνουμε αυτή την πρόταση είναι υπό ποιους κανόνες λειτουργεί ο συγκεκριμένος αγωγός. Ο χύψη ζέντα αγωγός. Όπως βλέπετε δεν έχει καμία σχέση αυτό με το ενεργειακό μείγμα και καμία σχέση φυσικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα που θέλουν να εξασφαλίσουν ορισμένα κράτη-μέλη. Τώρα, κάποιες άλλες ερωτήσεις που θα ήθελα να απαντήσω. Με τη σειρά που υποβλήθηκαν από τον κύριο Κάρεντ ήταν και ερώτηση του κύριου Μπούζεκ, νομίζω. Την ανάγκη για νέους κανόνες στους ισχύοντε αγωγού. Πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε διακρίσει ανάμεσα στου υπάρχοντε και νέους αγωγούς και γενικά υποδομές. Όταν κοιτάζετε την πρόταση επί της ουσίας, βλέπετε ότι δημιουργούμε ένα ελαφρύ εντό αγωγικών καθεστώ για τους ισχύοντες αγωγούς. Θέλουμε δηλαδή τα κράτη-μέλη να ψάξουν και να βρουν τι είναι απαραίτητο για να ευθυγραμμίσουν τους κανόνες που ισχύουν για τους ισχύοντες αγωγούς. Έχουμε προτείνει απλουστευμένες διαδικασίες για παρεκκλήσεις από κάποιες από τις αρχές, ούτως ώστε να λάβουμε υπόψη μας ότι αυτοί οι αγωγοί λειτουργούν ήδη. Και δεν θέλουμε φυσικά να δημιουργήσουμε βλάβη στη λειτουργία αυτών των αγωγών. Να δημιουργήσουμε πρόβλημα στη λειτουργία αυτών των αγωγών. Κύριος Κασνοντεύσκη, σας υπόσχομαι ότι η Κομισιόν θα παραμείνει στεναρεί με την πρόταση αυτή, γιατί πιστεύουμε σε αυτή την πρόταση, πιστεύουμε ότι είναι σωστή. Να σας υπενθυμίσω γιατί την προτείναμε κιόλα. Γιατί έγιναν πάρα πολλές συζητήσεις για το εφαρμοστέο δίκαιο και η Κομισιόν πάντα θεωρούσε ότι ακόμη και αν δεν έχουμε γραπτό δίκαιο, υπάρχουν κάποιοι άγραφοι νόμοι που ισχύουν και θα πρέπει να τους εφαρμόσουμε. Γιατί υπήρχαν νομικές διαμάχες στο παρελθόν και εμείς ξεκαθαρίσαμε ποιοι είναι οι κανόνες που ισχύουν τελικά. Είτε, κύριε Πίτερσεν, το ερώτημά σας για τις επιπτώσεις της τιμές φυσικού αερίου που θα έχει, επιπτώσεις που θα έχει η πρότασή μας. Μία σύντομη απάντηση. Και εσείς ο ίδιος είπατε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτή η αγωγή ε, να υπόκεινται στην πρόσβαση από την τρίτη χώρα, από το τρίτο μέρος. Αυτό θα αυξήσει τον ανταγωνισμό και θα μας βοηθήσει να έχουμε μια πιο ευρυθμή αγορά. Ο κύριος Ηλικιώτης έκανε τώρα μια άλλη ερώτηση και η κυρία Βέρνερ για τη μελέτη αντικτύπου. Έχετε δίκιο, κανονικά. Υπάρχει και εσωτερικός κανόνας. Συνοδεύουμε τις προτάσεις μας από μελέτη αντικτύπου. Γιατί πιστεύουμε ότι σε αυτήν την περίπτωση δεν χρειάζεται μια τέτοια μελέτη. Για το απλό γεγονός που ήδη ανέφερα, ότι για μα οι αρχές που τις ανέφερε και ο κύριος Πίτερσον, ε, ο διαχωρισμός, ε, δομή των τιμολογίων, πρόσβαση από τους τρίτους και διαφάνεια. Αυτές οι αρχές, με βάση τη δική μας νομική γνωμοδότηση, εφαρμόζονται ήδη. Επομένως, απλώς ξεκαθαρίζουμε το γεγονός αυτό έτσι περαιτέρω. Η Κομισιόν, λοιπόν, ακριβώ για αυτόν τον λόγο, μετά από σοβαρό προβληματισμό, κατέληξε το συμπέρασμα ότι για αυτή δικά την πρόταση δεν χρειάζεται μελέτη αντικτύπου, αλλά στηρίξαμε βεβαίως την πρότασή μας ε, πάνω σε ένα έγγραφο των υπηρεσιών μας, όπου αναφέρονται οι απαραίτητες πληροφορίες, όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Η σύγκρουση με το διεθνές δίκαιο. Μια άλλη ερώτηση. Και εδώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Δεν ισχυριζόμαστε με αυτή την πρόταση ότι ο, το δικό μας δίκαιο θα εφαρμόζεται και εξωεδαφικά, δηλαδή εκτός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφορά μόνο την ε, επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο εκεί ισχύει. Κυρία Βέρνερ, η νομική βάση είναι το άρθρο 194. Αν το διαβάσετε, βλέπετε ότι υπάρχουν δύο παραδείγματα γιατί αυτή η νομική βάση μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εμείς προωθούμε τον ανταγωνισμό με τη ρύθμιση της πρόσβασης των τρίτων, γιατί όπως είπα αυτό θα ενισχύσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας αυτό αναφέρει από τη 194 και η εφαρμογή της αρχής της διαφάνειας. Αυτό σημαίνει δημοσίευση των τεχνικών δεδομένων για τη λειτουργία αυτών των αγωγών. Και αυτό θα συνεισφέρει στην ασφάλεια ανεφοδιασμού. Ξέρουμε εκ των προτέρων τι γίνεται με αυτού του αγωγού. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό προφανώ θα αυξήσει την ασφάλεια. Κύριε Γιώργ, τελευταίο σημείο. Το πεδίο εφαρμογή. Πολύ συγκεκριμένη ερώτησή σα. Αυτή η πρόταση Εφαρμόζεται επίσης και σε αγωγούς που περνάνε από τη μια χώρα στην άλλη με χερσαίο τρόπο. Η Ουκρανία, η Ουγγαρία. Ναι, δεν αφορά μόνο τους υπεράκτιους αγωγούς, αλλά και τους χερσαίους αγωγούς που μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτη χώρα. Αυτά. Ελπίζω να απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις, Πρόεδρε. Ναι, έτσι νομίζω και εγώ. Λοιπόν, Κύριε Κάριν, ε, ξέρετε ότι εσείς πρέπει να πάρετε τώρα το λόγο για να συνοψίσετε. Αφού προβλέπετε, θέλετε να προσθέσει κάτι. Θα μιλήσω ως Γέρζι Μπούζεκ για άλλη μια φορά. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Ας συνεργαστούμε λοιπόν. Ωραία, εκτιμούμε πάρα πολύ τη σαφηνιά σας. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να καλωσορίσω τώρα τον κύριο Τίμπορ Ναυρατσίσα, τον Επίτροπο Αρμόδιο για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, την Νεολαία και τον Αθλητισμό, στα πλαίσια του διαρθρωμένου διαλόγου. Να σας πενθυμίσω ότι ο Επίτροπος Ναυρατσίσα προσκλήθηκε από την Επιτροπή μας στα πλαίσια του διαρθρωμένου αυτού διαλόγου μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο Επίτροπος θα μας ενημερώσει τώρα για την εφαρμογή του δικού του προγράμματος που έχει να κάνει με το πρόγραμμα εργασίας 2017 και θα μας πει πώς θα τα πράγματα του 2018. Κύριε Ναύρατσης, κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Βιομηχανίας, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με προσκαλέσατε να σας μιλήσω σήμερα το απόγευμα. Εκτιμώ ιδιαίτερα τη δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσω μαζί σας για τα επιτεύγματα, τις προκλήσεις και τη χάραξη πολιτικής τα ζητήματα πλέον πολιτικής δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ξεχωριστά και μονομένα. Σχεδόν κάθε θέμα απαιτεί πλέον συνεργασία διατομεακή σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Απαιτείται λοιπόν διαλλακτικότητα, ανοιχτό πνεύμα, πρέπει να παραμείνουμε σε γρήγορση, να ακούμε, να φουγκραζόμαστε τις άλλες απόψεις και να μπορούμε να συνεργαζόμαστε διατομεακά και διασυνοριακά. Το ανοιχτό αυτό πνεύμα, η διαλλακτικότητα αυτή απειλείται σήμερα. Εναπόκειται λοιπόν σε εμά να προασπίσουμε και να ενισχύσουμε τη διαλλακτικότητα αυτή και το ανοιχτό αυτό πνεύμα τώρα περισσότερο από ποτέ. Για να περιπλακούν περισσότερο τα πράγματα, η θέση των επιστημονικών αποδεκτικών στοιχείων τη σήμερα ημέρα απειλείται πάλι από μια πολλωμένη νοοτροπία που δεν νοιάζεται για τα περιστατωμένα επιστημονικά γεγονότα. Πρέπει και αυτό να το καταπολεμήσουμε. Μόλις συμμετείχα στην ετήσια διάσκεψη «Επιστήμη συναντά τα κοινοβούλια» στα πλαίσια του Κοινού Κέντρου Ερευνών και χαίρομαι πάρα πολύ που ήσασταν ορισμένοι από εσά εκεί και που συζητήσαμε μαζί πώς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη και γνώση υπέρ της χάραξης πολιτικών. Έχουμε καταβάλει σημαντικέ προσπάθειε προκειμένου η επιστημονική γνώση και οι περιστατωμένε επιστημονικέ αποδείξει να μπουν στο κέντρο τη χάραξη πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαφείται όλο και περισσότερο στο κοινό κέντρο ερευνών για την παροχή επιστημονικών συμβουλών και υποστήριξη σε σχέση με τι κοινοτικέ πολιτικέ. Το κοινό αυτό κέντρο ερευνών έχει αλλάξει πολύ τελευταία, μετασχηματίστηκε αποκτά πολύ πιο στρατηγικό ρόλο στη χάραξη πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και επικεντρώνεται σε ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Η αναδιοργάνωση του Κοινού Κέντρου Ερευνών του 2016 αποφέρει καπνούς, ε, καρπούς, με συγχωρείτε. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών πλέον γίνεται βασικός διαχειριστής της ε, γνώσης. Στα κέντρα γνώσης του Κοινού Κέντρου Ερευνών έχουμε πλέον εμπειρογνώμονες, καθώς επίσης και κέντρα αριστείας ε, εντό και εκτό Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Έχουμε κέντρα γνώσης πλέον στον τομέα τη διαχείριση κινδύνου από τι καταστροφέ, τη μετανάστευση και τη δημογραφία, στι εδαφικέ πολιτικέ και στη βιοοικονομία τα κέντρα αρμοδιότητα του κοινού κέντρου ερευνών χρησιμοποιούν πλέον εργαλεία ανάλυση όπω ανάπτυξη μοντέλων, δικτών, χρησιμοποιούν τη μέθοδο τη άντληση κειμένων καθώ επίση και μικροοικονομική αξιολόγηση. Αυτό εφαρμόζεται σε όλου του τομεί. Για παράδειγμα, το Κέντρο Αρμοδιότητας για τους σύνθετους δείκτες κατήρτισε τον πίνακα αποτελεσμάτων που ουσιαστικά παρακολουθεί την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Και σύντομα θα έχουμε και ένα κέντρο γνώσης όσον αφορά την απάτη στον τομέα των τροφίμων και την ποιότητα των τροφίμων. Η εμπειρογνωμοσύνη και η γνώση του Κοινού Κέντρου Ερευνών είναι στη διάθεση των κρατών μελών και είμαστε στη διάθεση των τοπικών και περιφερειακών αρχών επίση για να του παρέχουμε περισσότερε επιστημονικέ γνώσει. Αξιότιμα μέλη, η εργασία του Κοινού Κέντρου Ερευνών ανταποκρίνεται στι βασικέ προκλήσει που πρέπει να αντιμετωπίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι υπάρχει μια εξαιρετική συνεργασία με την εκσταστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τι μετρήσει εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία και σε ακροάσει που γίνουν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και στα πλαίσια του κοινού κέντρου ερευνών είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και χαίρομαι πάρα πολύ για την αντιπροσωπεία σα που ήρθε στην μονάδα του Ινστιτούτου Περιβαλλοντική Προστασία, στο ΙΣΠΡΑ. Αντιμετωπίζουμε στο πλαίσιο των κοινών κέντρων ερευνών πολλά πολύπλοκα ζητήματα. Για παράδειγμα, ζητήματα όπω η ουσία φιπρονίλη, γλυφοσάτη, ενδοκρινικοί διαταράκτε, οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, η η είναι όλοι κλάδοι δηλαδή τομεί επί τους οποίους το κοινό κέντρο ερευνών παρέχει εγκαίρω επιστημονικά δεδομένα. Επίση, χρησιμοποιήθηκε η εμπειρογνωμοσύνη του κοινού κέντρου ερευνών προκειμένου να καταφέρουμε να καταλήξουμε στην συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και συνεργάζεται το Κοινό Κέντρο Ερευνών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γενικότερα για τι δικλείδε ασφάλεια και γενικότερα την ασφάλεια στον τομέα τη πυρηνική ε, ενέργεια. Προσπαθούμε όμω να ασχοληθούμε και με τεχνική νοημοσύνη και τα μαζικά δεδομένα. Σε έναν όλο και πιο στεδεμένο κόσμο και ένα όλο πιο πολύπλοκο κόσμο χρειαζόμαστε καινοτόμου τρόπου προσέγγιση και επίλυση των προβλημάτων. Η σχέση μεταξύ επιστήμη, πολιτική κοινωνία δεν είναι ούτε ξεκάθαρη ούτε γραμμική. Πρέπει λοιπόν να προσαρμόσουμε την μέθοδο λήψη αποφάσεών μα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τι νέε κοινωνικέ και τεχνολογικέ προκλήσει. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη Γνώση του Κέντρου Ερευνών και θα ήθελα πραγματικά να σα καλωσορίσω για μια ακόμα φορά στι μονάδε που έχουμε, τι ερευνητικέ τη Ίσπρα, στο Πέτεν, στο Γκέλ, στην Καλστρούη και στη Σεβίλη αξιότιμα μέλη. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομία και Τεχνολογία, καθώ επίση και στι δράσει Μαρή Κλοντόφσκα Κιουρί, που συμβάλλουν και τα δύο πάρα πολύ σημαντικά στην καινοτομία, την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, επενδύοντα στι δεξιότητε και τι αρμοδιότητε των πολιτών. Η ενδιάμεση αναθεώρηση του Ορίστου 2020 καταδεικνύει ότι το μοντέλο EAT για την καινοτομία λειτουργεί σωστά και ενσωματώνει την εκπαίδευση, την έρευνα και την επιχειρηματικότητα σε μακροχρόνιες εταιρικέ σχέσει που εμπλέκουν τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα η κοινότητα EIT απευθύνεται σε χίλιου περίπου εταίρου εντό και εκτό τη Ευρώπη. Έχουμε έξι κοινότητε γνώση και κοινοτομία που ήδη λειτουργούν και δύο ακόμα θα ξεκινήσουν το έργο του του χρόνου. Και πάνω από 40 κέντρα συστέγαση αυτή τη στιγμή αντιμετωπίσουν σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις στις περιφέρειές σας. Οι απόφοιτοι του Ινστιτούτου του EIT έχουν καλύτερες πιθανότητες έβρασης μιας καλής θέσης εργασίας και έχουν περισσότερες, υψηλότερους μισθούς από άλλους πτυχιούχους. Επίσης συμβάλλουμε πάρα πολύ στο να υποστηρίξουμε χρηματοδοτικά νεοφυείς επιχειρήσεις. Φέτος το περιοδικό Forbes συμπερίλαβε 18 αποφύτους του EIT στον κατάλογο 30 κάτω των 30 με του επιφανέστερου νέους επιχειρηματίες, εφευρέτες καινοτόμους και επιστήμονε με σημαντική επιρροή. Πρέπει να είμαστε λοιπόν περήφανοι για τα όσα έχουμε πετύχει και να είμαστε φιλόδοξοι για το μέλλον. Πρέπει να ενισχύσουμε και να βαθμίσουμε τι εκπαιδευτικέ μα δραστηριότητε, ιδίω αυτέ που φέρουν τη σήμανση EIT, που θα πρέπει να γίνει πραγματικά το σήμα κατεθέν τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την επιχειρηματική εκπαίδευση. Και θα πρέπει να αυξήσουμε επίση τον περιφερειακό αντίκτυπο μέσω των κοινών αυτών κέντρων ερευνητική συστέγαση. Δεν θα πρέπει καμία περιφέρεια να μείνει πίσω και ιδίω να βοηθήσουμε αυτέ οι οποίε υπολείπονται και καθυστερούν αυτή τη στιγμή. Το Ινστιτούτο αυτό έχει δείξει ήδη την ικανότητά του να καταφέρει να προσαρμόζεται και να εξελίσσεται, μολονότι παραμένει πάρα πολύ σταθερό στα βασικά στατικά του στοιχεία. Επενδύσει στον ανθρώπινο παράγοντα για την καινοτομία και για να αντιμετωπίσουμε κοινωνικά προβλήματα. Καθώ προχωράμε στο νέο ερευνητικό πρόγραμμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιμείνουμε σε αυτά τα στοιχεία. Ολοκληρώνοντα, θα ήθελα να πω κάποια λόγια για τι δράσει Μαρή Λοντόφσκα Κιουρί. Φέτο γιορτάζουμε την 20η επέτειο από τη θέσπιση του προγράμματο Μαρή Λοτόφσκα Κιουρί που έχει υποστηρίξει χρηματοδοτικά 100.000 ιδιαίτερα ταλαντούχους ερευνητές ενισχύοντας τις δεξιότητές τους και δίνοντα νέα όθηση στην επαγγελματική του σταδιοδρομία. Ορισμένοι από του επιστήμονε αυτού συνέβαλαν σε πρωτοποριακέ έρευνε και αναγνωρίστηκαν ή βραβεύτηκαν φέτο με τα βραβεία Νόμπελ Φυσική και Χημία. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που διοργάνωσε την εκδήλωση Science is Wonderful, επιστήμη είναι καταπληκτική, πέρυσι το Σεπτέμβριο, το τελευταίο μάλλον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για μια σημαντική εκδήλωση η οποία οδήγησε στη βραδιά Ευρωπαίων ερευνητών όπου συμμετείχαν περίπου ένα εκατομμύριο πολίτε σε εκδηλώσει που γίνανε σε περίπου 340 πόλει Ευρωπαϊκή Ένωση Να ευχαριστήσω επίσης την Επιτροπή σας γιατί τονίσατε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές επιτυχίες των δράσεων Μαρίς Λοντόφσκα Κιουρί. Και να ευχαριστήσω επίσης την Σολεδάδ Καπεθόν Ριθ, την εισηγήτριά σα, για το ζήτημα αυτό. Θα ήθελα πραγματικά η Ευρώπη να γίνει ένα ηγετικό κόμβο για τη νέα γενιά παγκόσμιων ταλέντων. Και οι δράσει Μαρή Λοντόφσκα Κιουρίδη δραματίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Για παράδειγμα, θα πρέπει να δούμε πώ μπορούμε να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τι ανάγκε των κρατών μελών που παρουσιάζουν αυτή τη στιγμή καθυστέρηση, χωρί όμω να υπονομεύουμε τη βασική αρχή τη αριστεία. Ήδη έχω λάβει δράση δεσμεύοντα 18 εκατομμύρια ευρώ για τα, επόμενα, για τα τελευταία μάλλον τρία χρόνια του προγράμματος ορίζοντας 2020 προκειμένου να χρηματοδοτηθούν περισσότερες υποτροφίες. Κατά αυτόν τον τρόπο περισσότερες χώρες και περισσότεροι ερευνητέ θα μπορούν να υποφεληθούν από τη χρηματοδότηση αυτή, ιδίως όσοι δεν κατάφεραν να έχουν πρόσβαση στις υποτροφίες Marie Curie. Πρέπει να προωθήσουμε νέες μορφές αριστείας. Χαίρομαι πάρα πολύ που ένα 40% των υποτρόφων των δράσεων Marie Curie είναι γυναίκες, αλλά μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Έχουμε διπλασιάσει αυτή τη στιγμή τον προπολογισμό για τις γυναίκες εκείνες που επιστρέφουν στον τομέα της έρευνας αφού κάνανε ένα σύντομο διάλειμμα στην επαγγελματική του σταδιοδρομία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει κατάληξη ισορρόπηση, μια ισορροπημένη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στα ερευνητικά προγράμματα. Το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για λόγου δικαιοσύνη, αλλά γιατί προωθεί την αριστεία και διατηρεί την Ευρώπη στην αιχμή του δόρατο όσον αφορά την έρευνα. Αξιότιμα μέλη, Πιστεύω ότι ε, έδειξε την αποφασιστικότητά μου όσον αφορά τα αποτελέσματα τα οποία πρέπει να προωθήσουμε στον τομέα τη επιστήμη, τη έρευνα, τη εκπαίδευση και τη οικονομία. Εξέφρασα τι απόψει μου και περιμένω τώρα και τι δικέ σα ερωτήσει. Ευχαριστώ πολύ. Επίτροπε, από τι διάφορε πολιτικέ ομάδε, οι διάφοροι μιλητέ. Ο κύριο Κάρεντ δεν είναι παρόν. Μήπω θα θέλει ο κύριο Λεβαντόφσκι να πει κάτι. Θα σας εκπλήξω. Σας ευχαριστώ, Επίτροπε, για την παρουσία σας. Ε, καλό σημάδι. Μία σύντομη παρουσίαση. Σας ευχαριστώ που προφέρατε και τόσο εύκολα και τόσο σωστά ε, το πρόγραμμα αυτό, που είναι το πιο σημαντικό πρόγραμμα για νέους ερευνητές. Μαρή Σκλοντόφσκα Κιουρί. Είναι η μόνη γυναίκα η οποία έχει πάρει ε, βραβείο Νόμπελ στην ιστορία. Ο κύριος Καρνοντεύσκη δεν είναι εδώ. Ο κύριος Τσέσσαρ, όχι. Ο κύριος ε, Πίτερσον εκπροσωπεί τον κύριο Φέντερ Θέλει να πει κάτι. Παρακαλώ. Γνέφω εδώ πέρα, σηκώντα το καρτελάκι, αλλά δεν με βλέπετε. Ευχαριστώ για την παρουσίαση, Επίτροπε. Ενδιαφέρουσα. Μία σύντομη ερώτηση. Για την ιατρική έρευνα, κάνετε κάτι. Στην Ίσπρα γίνεται τίποτα για τα απόβλητα στους ωκεανούς ε, και μια και μας περιβάλλει το νερό, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε κάτι και για τη θάλασσα και τους ωκεανού. Ε, κάντε κάτι στην Ίσπρα για τους ωκεανού και τα απόβλητα στου ωκεανού. Ο κύριος Κούλιτσεκ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, δυστυχώ ε, δεν μιλούμε ουγγρικά σήμερα. Ε, ζητώ συγγνώμη, δεν, μιλώ εγώ ουγγρικά. Ε, έχω ένα ερώτημα. Ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ασχολείται με ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, μια τεράστια πρόκληση. Πώς θα προχωρήσουμε σε μια αποτελεσματική ε, εκπαίδευση, ένταξη των μεταναστών στην εκπαίδευση. Ε, υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις ε, στη, Γερμανία η καγκελάριος λέει θα τα καταφέρουμε στη Σουηδία υπάρχουν 60 πλέον ζω, ζώνες στις οποίες δεν έχει πρόσβαση η αστυνομία και εμείς δυστυχώς έχουμε αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα χιλιάδων ανθρώπων οι οποίοι ούτε θέλουν ούτε μπορούν ε, στην πραγματικότητα να εκπαιδευτούν και να κάνουν οποιαδήποτε πρόοδο. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους Ρωμά. Ε, με ενδιαφέρει λοιπόν να μου πείτε ως ε, ε, ως πολιτικό υπεύθυνο που κι εσείς μαζί με άλλους φέρατε όλους αυτούς τους χιλιάδες πρόσφυγες στην Ευρώπη. Ε, πώς θα καταφέρουμε όλοι αυτοί οι άνθρωποι να ενταχθούν στις κοινωνίες μας, να μάθουν τις γλώσσες μας, τις νοοτροπίες μας, τα ήθη μας, τα ήθημά μας, που είναι και διαφορετικά σε κάθε χώρα βέβαια. Ε, πώς ακριβώς λοιπόν σκοπεύετε εσείς να υποστηρίξετε τις επιμέρους δράσεις και προσπάθειες των κρατών μελών. Όχι φυσικά να στείλουμε τους ανθρώπους αυτούς ε, σε εγκαταλελειμμένα χωριά. Θέλω να μου πείτε πώς ακριβώς φαντάζεστε ότι οι άνθρωποι αυτοί θα καταφέρουν κάποια στιγμή στο μέλλον να ζήσουν με βάση τις ε, ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τα πρότυπα. Ευχαριστώ κύριε Κότσεκ. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις ή σχόλια, παρεμβάσεις. Όχι. Οπότε θα ήθελα να ζητήσω από τον Επίτροπο Νάβασες να απαντήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά τις δραστηριότητες του Κοινού Κέντρου Ερευνών, φυσικά και το Κοινό Κέντρο Ερευνών ε, έχει ερευνητικά ενδιαφέροντα στον τομέα της ιατρικής και, και στην Ίσπρα, στη μονάδα μας στην Ίσπρα. Υπάρχει μάλιστα και μια μονάδα ε, συγχώνευσης και συγκέντρωσης δεδομένων και στατιστικών στοιχείων ε, για τον ε, καρκίνο, τον επιπολασμό της ασθένειας αυτής. Επίσης ασχολούμαστε πολύ με ζητήματα θαλάσσιας ε, ρήπανσης, ρήπανσης των ωκεανών Υπάρχει άλλωστε και αρμόδιο επίτροπο, με τον οποίο βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή και συνεργασία για αυτά τα θέματα. Όσον αφορά το ζήτημα τη μετανάστευση κοινωνική ένταξη των Ρωμά και όλων των υπόλοιπων πληθυσμιακών ομάδων. Νομίζω ότι αυτό το θέμα υπερβαίνει τις δικές μας ε, αρμοδιότητες. Το Κοινό Κέντρο Έρευνας ε, έχει βεβαίως γνώσεις και στον τομέα της μετανάστευσης και στον τομέα της αντιμετώπισης ε, καταστροφών. Ε, που αυτές οι καταστροφές άλλοτε είναι φυσικές, άλλοτε είναι και κοινωνικές. Υπάρχουν λοιπόν αυτές, αυτά τα κέντρα γνώσεων που είναι κέντρα αριστείας, εμπειρογνωμοσύνη, όπου συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με επιτυχημένες ε, στρατηγικές αντιμετώπισης των ριζικών αιτίων αυτών των φαινομένων, όπου ακριβώς μέσω αυτών των κέντρων τίθεται στη διάθεση όλων των κρατών μελών ε, όλη αυτή η γνώση που έχει συγκεντρωθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και πέρα από το JRC στο δικό μου χαρτοφυλάκιο βεβαίως εντάσσεται και το πρόγραμμα Erasmus το οποίο δεν αφορά βεβαίω μόνο την κινητικότητα των φοιτητών. Κατά κύριο λόγο βέβαια αφορά την κινητικότητα των, των φοιτητών, αλλά περιλαμβάνει και ορισμένε άλλε δράσει όπω εκμάθηση γλωσσών. Ε, υπάρχει στο, στο πλαίσιο του προγράμματο αυτό συνεργασία με μη κυβερνητικέ οργανώσει οι οποίε ασχολούνται με, το θέμα, με τα θέματα κοινωνική ένταξη, Ρωμά αλλά και άλλων ομάδων μεταναστών. Και την προηγούμενη εβδομάδα μάλιστα ε, απένιμα για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Βραβείο Κοινωνικής Ένταξης μέσω του αθλητισμού μέσω του οποίου αναγνωρίζεται η δράση και η συνεισφορά εκείνων των μη κυβερνητικών οργανώσεων που ξεκίνησαν ε, χρήσιμα προγράμματα ε, στις τοπικές κοινωνίες για την ένταξη ε, νεοαφιχθέντων μεταναστών μέσω ε, του αθλητισμού. Έχουμε λοιπόν μια ολόκληρη πλειάδα, μια ολόκληρη γκάμα εργαλείων και μέσων μέσω των οποίων υποστηρίζουμε τις δράσεις κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο. Ευχαριστώ κύριε Ναύρατσης. Επειδή έχουμε λίγο χρόνο μέχρι να ξεκινήσουμε τη συζήτηση του επόμενου θέματος, θα ήθελα ε, να προσθέσω ένα τελευταίο ερώτημα. Ένα ερώτημα που θα περιμένατε να το λάβετε από κάποιον, κάποιο μέλος της ομάδας ECR. Το ερώτημα είναι γιατί χρειαζόμαστε Επίτροπο Παιδείας. Στην ε, δική μου χώρα η παιδεία είναι αρμοδιότητα των ε, κρατηδίων και τα κρατήδια της Γερμανίας διατηρούν πάντοτε την, ε, την, την αρμοδιότητα αυτή, ότι εκείνα είναι υπεύθυνα για την παιδεία. Τι θα τους πω, πώς μπορώ να, να δικαιολογήσω την ύπαρξη ενός επιτρόπου παιδείας, ε, ο οποίος έχει περισσότερες αρμοδιότητες πέραν από το ε, Erasmus+. Φαντάζομαι ότι ξέρουν τα, οι εκπρόσωποι των κρατηδίων της Γερμανίας ότι υπάρχω και ότι βρίσκομαι ε, εδώ στην Επιτροπή σας. Σύμφωνα με την ε, συνθήκη, ο ρόλος, μας, ο ρόλος μου είναι να προσθέσω μια ευρωπαϊκή διάσταση και ευρωπαϊκή προστεθέμενη αξία στην, ε, στην παιδεία. Μετά τη διάσκεψη των Παρισίων το 2015 υπήρξε ένα ε, έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας, όπου οι Υπουργοί Παιδείας των κρατών μελών και εγώ ε, προχωρήσαμε στην ε, διακήρυξη των Παρισίων, όπου αποσαφηνίζονται οι βασικοί στόχοι και ο ρόλος των εκπαιδευτικών συστημάτων στην, στην, όσον αφορά την συμμετοχή στο δημοκρατικό πολίτευμα των νέων πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό ε, διοργανώνονται και ε, διάφορα εργαστήρια και σεμινάρια με τη συμμετοχή νέων ανθρώπων από όλη την Ευρώπη όπου εξετάζονται ζητήματα ε, που άπτονται του κοινωνικού ρόλου των εκπαιδευτικών συστημάτων πώς τα εκπαιδευτικά συστήματα μπορούν να συμβάλλουν και να βοηθήσουν την κοινωνία ώστε να διαπαιδαγωγούνται υπεύθυνοι όρεμοι πολίτες σε μια δημοκρατική κοινωνία ε, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο και το πρόβλημα της ριζοσπαστικοποίησης και ένα άλλο ε, ε, παράδειγμα είναι βεβαίως οι δραστηριότητες σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πρόσφατα υιοθετήσαμε, εγκρίναμε την σχετική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση που παρέχει κατευθυντήριες γραμμές σε εκείνα τα κράτη-μέλη που θέλουν να επιτύχουν νέους υψηλότερους στόχους για τα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τους. Για παράδειγμα, ένα, μία από τις διαπιστώσεις μας τα τελευταία χρόνια είναι ότι τα πανεπιστήμια δεν ε, αρκεί να είναι απλά χώροι ε, μεταλαμπάδευσης ε, και παράδοσης γνώσης αλλά θα πρέπει ενεργά να συμμετέχουν και στη ζωή ε, κοινωνική, οικονομική ε, των τοπικών ε, κοινωνιών, να βοηθούν δηλαδή στην αναζωογόνηση των κοινωνικών δραστηριοτήτων αλλά και της οικονομικής δραστηριότητας σε τοπικό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ, λέω Προεδρεύων, και περνάμε στο επόμενο θέμα της σημερινής διάταξής μας που είναι ο Acer. Θα υπάρξει μια... Ε, παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης παρακολούθησης της αγοράς και ανταλλαγή απόψεων με τον διευθυντή του Acer, τον κύριο Ποτότσνικ. Ο, κύριε Ποτότσνικ, αν δεν έχετε αντίρρηση, σας καλώ να ανέβετε εδώ στο βήμα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για την παρουσία σας. Και μια και είμαι ε, σκιώδης εισηγητής της ομάδας μου για αυτό το θέμα, πρέπει να σας πω ότι έχω ήδη συναντηθεί με τον κύριο Ποτότσνικ. Ε, δεν νομίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Κύριε Ποτότσνικ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να σας ζητήσω συγγνώμη Ο Λόρτ Mog ε, έρχεται, είναι καθοδόν. Πρέπει να σας πω ότι δεν είναι πλέον πρόεδρος ε, του Συμβουλίου Ρυθμιστικών Αρχών. Ο κύριος Μπλάνι ε, ορίστηκε πρόεδρος, εξελέγει και ορίστηκε πρόεδρος τον προηγούμενο μήνα. Παρ' όλα αυτά αποφασίσαμε ο Lord Mog ε, να κάνει μαζί μου αυτήν την παρουσίαση. Πρώτον, να σας πω ότι η παρουσίαση αυτή θα είναι συντομότερη από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Καλό θα είναι αυτό για να μπορείτε να θέσετε και τα ερωτήματά σας. Όπως είναι και η έκθεση μικρότερη σε έκταση. Και αυτό οφείλεται μεταξύ άλλων στο γεγονό ότι ο προπολογισμό μα μειώθηκε κατά 16%, γι' αυτό και χρειάστηκε να σφίξουμε κάπως τα ζωνάρια και να επικεντρωθούμε στα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία ε, όσον αφορά την ε, εξέλιξη της εσωτερικής αγοράς. Ε, επικεντρωθήκαμε λιγότερο στο ζήτημα του λιανικού εμπορίου, αν και σήμερα πρέπει να σας πω ότι ανακοινώθηκε ότι υπάρχει μια σχετική μελέτη που επικεντρώνεται συγκεκριμένα στο ελληνικό επίπεδο. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω την, την ε, Επιτροπή Ήτρε, την Επιτροπή Προπολογισμών, ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για, το, για την υποστήριξή τους ε, όσον αφορά τους δημοσιονομικούς περιορισμούς που ε, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε η Ολομέλεια μας υποστήριξε, δυστυχώς όμως στον τριμερή διάλογο τελικά δεν καταφέραμε να είμαστε μεταξύ εκείνων των οργανισμών που ε, είχαν προτεραιότητα όσον αφορά την χρηματοδότησή τους. Έτσι λοιπόν είμαστε ε, από τους οργανισμούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω μειωμένου προϋπολογισμού. Λοιπόν, τα βασικά ε, πορίσματα της, της, μελ, της μελέτης ε, αφορούν ε, την, το χοντρεμπόριο, ε, την, το λιανεμπόριο και την προστασία των καταναλωτών. Και νομίζω ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία, θετικά μηνύματα. Ας δούμε εδώ την αγορά φυσικού αερίου, ιδίως την, την αγορά. Βλέπετε εδώ ότι το κόστος ανεφοδεσμού ε, έχει μειωθεί. Ο, η τιμή λοιπόν ε, του τελικού καταναλωτή ε, είναι χαμηλότερη. Βλέπετε εδώ με κίτρινο το TTF, τον κόμβο ε, των κάτω χωρών ως αναφορά και με κίτρινο χρώμα είναι οι χώρες που πληρώνουν λιγότερο από ένα ευρώ με ανοιχτό μπλε ε, χώρε που πληρώνουν 1 έω 3 ευρώ και με σκούρο μπλε ε, χώρε που πληρώνουν πάνω από 3 ευρώ. Βλέπετε λοιπόν ότι τα τελευταία χρόνια ε, η κίτρινη περιοχή Ευρώπη Ευρώπης διευρύνεται. Και αυτό που είναι ενδιαφέρον τουλάχιστον από τη δική μου σκοπιά, είναι ότι η κίτρινη περιοχή διευρύνεται από, από το κέντρο της Ευρώπης προς τα, προς τις, προς τα άκρα. Ε, θα περίμενε κανείς ότι το φυσικό αέριο θα ήταν πιο φθηνό ε, όσο πιο κοντά πάμε στην, ε, στην, στην πηγή Δεδομένου λοιπόν ότι το φυσικό αέριο προέρχεται από την Ανατολή της, ε, της Ευρώπης, θα περίμενε κανείς ότι εκεί θα ήταν πιο φθηνό. Δεν συμβαίνει όμως κάτι τέτοιο. Βλέπετε το κίτρινο, ε, τελικά ότι η τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής για το φυσικό αέριο ε, καθορίζεται από μια σειρά από παράγοντες, ανταγωνιστικότητα, υποδομές κτλ. Και σε αυτό τον τομέα έχουμε δώσει μεγάλη σημασία, ακριβώς γιατί τέτοιες ήταν και οι προσπάθειες που δόθηκαν στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς. Βλέπουμε λοιπόν μια μεικτή ε, εικόνα, αν δείτε την ε, απόδοση ε, διαφόρων κόμβων φυσικού αερίου και τους ταξινομήσαμε με βάση ορισμένους δείκτες. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι υπάρχουν κάποιοι ε, καθιερωμένοι κόμβοι, TTF, και το Εθνικό Σημείο εξισορρόπηση στην Ευρωπαϊ... στην... Ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχουν όμω και κάποια άλλη στοιχεία. Πάντως θετικό στοιχείο από πέρσι είναι ότι τόσο ε, ο Σλοβακικό όσο και ο τσεχικό κόμβο κατάφεραν και ανέβηκαν μια βαθμίδα στην κλίμακα και ανέβηκαν κατηγορία δηλαδή. Βλέπουμε λοιπόν ότι και σε εθνικό επίπεδο υπάρχει κινητικότητα, όχι μόνο ω προ την ολοκλήρωση ε, των αγορών, αλλά και όσον αφορά την απόδοση των κόμβων σε ολόκληρη την Ευρώπη να ε, στραφώ τώρα στο θέμα της ε, ε, ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό τον, τον χάρη τον έχετε δει πολλές φορές με διάφορα χρώματα και διάφορες αποχρώσεις. Εδώ βλέπετε την εδώ ε, βλέπετε με κόκκινο τη διασύνδεση των αγορών. Ε, με όλα τα χρώματα, όχι μόνο με το, με το κόκκινο. Καταγράφουμε το επίπεδο διασύνδεση των αγορών, σε ποιο βαθμό δηλαδή ε, είναι διασυνδεδεμένε οι ευρωπαϊκέ αγορέ. Αυτή τη στιγμή έχουμε τις διασυνδεδεμέ... μια διασυνδεδεμένη αγορά μεγάλη, μια περιοχή από το Γιβραλτέρ μέχρι την, ε, την θάλασσα του. Ε, υπάρχει, με μπλε περιοχή, υπάρχει μια κόκκινη περιοχή όπου συμμετέχουν τέσσερις χώρες. Έχουμε αυτή τη στιγμή 46 ε, ε, σύνορα στην Ευρώπη, τα οποία είναι διασυνδεδεμένα. Συν τρι, τρεις χώρες και υπάρχουν ακόμα 12 ε, χώρες διασύνδεσης που ακόμη λείπουν. Στόχο μας είναι λοιπόν να ολοκληρωθεί η διασύνδεση ολόκληρης της Ευρώπης στο συντομότερο δυνατό. Γιατί τα κάνουμε αυτό. Διότι αν δεν υπάρχει αυτή η διασύνδεση, η ηλεκτρική ενέργεια κινείται προς την, προς την λάθος κατεύθυνση και το έχουμε εξηγήσει σε παλιότερες ε, συζητήσεις μας. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει ε, και μικρότερη αποτελεσματικότητα στην λειτουργία των αγορών. Βλέπετε... Ε, ότι πριν από έξι χρόνια όταν ξεκινήσαμε τις μετρήσεις υπήρχε μια ε, αποδοτικότητα 86%. Την έχουμε όμως αυξήσει και βελτιώσει αυτή την αποδοτικότητα. Τι εννοώ με, τον όρο αποδοτικότητα. Να εξασφαλίζουμε ότι η ενέργεια ε, κινείται και κυκλοφορεί προς τη σωστή κατεύθυνση όποτε κρίνεται αναγκαίο με βάση τις τιμές ε, ή για περιβαλλοντικούς λόγους. Αν δείτε την μελέτη θα, θα διαπιστώσετε ότι σε μια σειρά από ε, συνοριακά σημεία η ηλεκτρική ενέργεια ε, ρέει προς την ε, λάθος κατεύθυνση. Είναι εκείνα τα σημεία όπου δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η διασύνδεση. Κατά τη, διάρκεια της ημέρας υπάρχει πάντοτε υπάρχει μια διακύμανση. Έχουμε φτάσει μόνο, μόνο έως το 50% και στην εξισορρόπηση ε, επίσης ε, ε, απομένουν ακόμα πολλά να γίνουν για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση στην αγορά το ευρωπαϊκό σύστημα διασύνδεσης αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή την επόμενη χρονιά και αναμένεται να ενισχυθεί και να βελτιωθεί πολύ η αποδοτικότητα του συστήματός μας. Ε, το ίδιο βεβαίως ε, και η εξισορρόπηση, η δυνατότητα της εξισορρόπησης της αγοράς. Αυτά είναι τα θετικά μηνύματα που σας φέρνω. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη σοβαρές προκλήσεις που δεν έχουμε αντιμετωπίσει. Η βασική πρόκληση που αυτή τη στιγμή ε, έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει είναι όσον αφορά η ικανότητα που διατίθεται προς εμπορική συναλλαγή. Πώς, πώς η ικανότητα δηλαδή τίθεται στο εμπόριο. Το πακέτο μέτρων που είχαμε προτείνει ε, πρόσφατα ε, προέβλεπε την οικοδόμηση διαφόρων έργων και προγραμμάτων ε, μέσω συμπράξεων και συνεργειών. Και πολλές υποδομές χρειάζονται ακόμη. Πολλά μπορούν όμως να γίνουν ε, και με την αξιοποίηση της υπάρχουσας ε, υποδομής που υπάρχει στην Ευρώπη. Και εδώ σε αυτό, τον, σε αυτό το γράφημα βλέπετε σε ποιο βαθμό οι υποδομές που υπάρχουν ήδη αυτή τη στιγμή αξιοποιούνται για, την, για τις εμπορικές συναλλαγές. Αυτή λοιπόν είναι η ικανότητα δίκτυ, η συγκριτική ικανότητα να το πω έτσι, πόσο θα μπορούσαν δηλαδή να αξιοποιηθούν οι υποδομές. Κατά μέσο όρο, μόλις ε, οι υποδομές στην Ευρώπη ε, αξιοποιούνται μόνο για το 50% της διάθεσης των ε, ε υπαρχών των ποσοστήτων ενέργειας στην αγορά. Υπάρχουν κάποιες περιφερειακές αλλαγές βεβαίως, αλλά βλέπετε ότι στην νοτιοανατολική Ευρώπη μόλις το 1 τέταρτο ή το 1 πέμπτο ε, της ποσότητας ενέργειας που θα μπορούσε να τεθεί σε εμπορική διάθεση τελικά τίθεται ε, ε, στο εμπόριο. Και αυτό είναι μια πρόκληση, γιατί αυτή που αυτό είναι μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Πέρσι είχαμε μάλιστα δημοσιεύσει μια σύσταση προκειμένου να αποφύγουμε κάποιε ακραίε καταστάσει τι οποίε αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή ανάμεσα στη Γερμανία και στο Πολωνία η διαθέσιμη ικανότητα ήταν σχεδόν 0% ενώ τιμέ τιμές ε, καταγράφηκαν και σε πολλά άλλα συνοριακά σημεία. Ε, μιλάμε για ένα πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο ποσοτήτων ενέργεια που διατίθεται στην αγορά. Ε, Τσεχία-Πολωνία 1%, Σλοβακία-Πολωνία 2% ε, και σε άλλα συνοριακά σημεία βλέπετε ότι ε, κινείται γύρω στο 10-15%. Και αυτό σχετίζεται πάντοτε με τον υπολογισμό των ικανοτήτων. Και εμεί θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν αλλαγέ ή διακρίσει ανάμεσα στι εσωτερικέ και τι διασυνοριακέ ανταλλαγέ. Ε, αυτό βεβαίως έχει και ιστορικό χαρακτήρα, πώς είχαν χτιστεί και πώς είχαν ε, διαμορφωθεί ε, αυτά τα συστήματα στο παρελθόν. Θέλουμε όμως πλέον να υπερβούμε τα, τα, τα εμπόδια του παρελθόντος για να δημιουργήσουμε μια πραγματική ενιαία αγορά και να κινηθούμε μακριά από αυτή την παλιά παροχημένη ε, προσέγγιση. Βεβαίως δεν περιμένουμε ότι η εφαρμογή της σύστασής μας θα έχει δραματικές ε, επιπτώσεις, θα επιφέρει δραματικές αλλαγές, αλλά τουλάχιστον αυτό που σκοπεύουμε, ε, αυτό που, στο οποίο αποσκοπούμε είναι να αλλάξουμε νοοτροπία, να υπάρξει μια αλλαγή του υποδείγματος βάσει του οποίου προσανατολίζονται οι εθνικές αρχές και οι επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που η Κομισιόν έλαβε υπόψη της δύο από τις συστάσεις μας στο χειμερινό πακέτο της και θα παρέχουμε κάθε βοήθεια στην Κομισιόν προκειμένου να εφαρμοστούν αυτές οι συστάσεις μας διότι ε, είναι πραγματικά κρίσιμη σημασία οι υπάρχουσες υποδομές να ε, αξιοποιούνται ε, στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Φυσικά όλα αυτά απαιτούν χρόνο ε, αν και με τη δική μας βοήθεια ε, θεωρούμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάποια βήματα πιο γρήγορα από ό,τι μέχρι τώρα. Λοιπόν, για να επανέλθω στα καλά μηνύματα. Φέτος, για πρώτη φορά, βλέπουμε τα επιτεύγματα στο, στην ε, αγορά χονδρικής και την ε, τελική κατα, τιμή καταναλωτή. Κάθε χρόνο βλέπαμε ότι υπήρχαν κάποιες θετικέ εξελίξεις στην αγορά χοντρική, χωρίς όμως να ωφελούνται οι καταναλωτές. Φέτος όμως βλέπουμε ότι τόσο οι επιχειρήσεις όσο και τα νοικοκυριά άρχισαν να υποφελούνται από τις χαμηλότερες τιμές στην αγορά χοντρική. Πλέον δηλαδή ε, μετακυλίεται αυτό το όφελο στο οικονομικό και στον τελικό καταναλωτή. Μέχρι στιγμής Αυτά τα ωφέλη στη χανδρική αγορά αντισταθμίζονταν από, την, από τις χρεώσεις για την υποστήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πλέον όμως ε, υπάρχει πραγματική μείωση στην, ε, στην, στις τιμές καταναλωτή. Επίσης, σε επίπεδο λιανικής αγοράς ε, κοιτάξαμε τι ακριβώς τελικά πληρώνουν οι καταναλωτέ και σε ποιο βαθμό ο ανταγωνισμός μπορεί να αναπτυχθεί και να διευρυνθεί στο επίπεδο της λιανική αγοράς. Εδώ τα πράγματα ε, ε, ε, παρουσιάζουν πολύ μεγάλη ποικιλία, ποικιλομορφία. Πράγματι, οι τιμέ καταναλωτή μειώνονται, ωστόσο η αναλογία του τι πληρώνει ο κάθε, ο κάθε καταναλωτής, ένα στοιχείο που είναι ανοιχτό στον ανταγωνισμό, επίση ποικίλει σοβαρά πολλές φορές η τιμή δεν, ε, ε, ε, δεν καθορίζεται μόνο ή κυρίως από την, από την τιμή του εμπορεύματος αλλά από διάφορες άλλες χρεώσεις που επιβάλλονται στους καταναλωτές. Άρα ο ανταγωνισμός, το κομμάτι στο οποίο υπάρχει ανταγωνισμός συμπιέζεται στον τελικό λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Βλέπετε εδώ λοιπόν ότι οι προμηθευτές μπορούν να ανταγωνίζονται σε ένα περιθώριο 35 cent για κάθε ευρώ που καταβάλλεται ως τιμή. Και έτσι λοιπόν ε, ε, πολλές φορές ε, τελικά θολώνεται η εικόνα του τι πληρώνει ο καταναλωτές λόγω των πολλών, πολλαπλών χρεώσεων που επιβάλλονται σε αυτόν μέσω των, των λογαριασμών σε αυτόν άλλων τελών και χρεώσεων όπως είπα κάποια από αυτά τα, χρέη, από αυτά τα τέλη, μάλλον πολλές, από αυτές τις χρεώσεις ε, δεν συνδέονται ή συνδέονται ελάχιστα με το, με το, με το κατεξοχήν εμπόρευμα δηλαδή του, της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτά, εν πάση περιπτώσει, ως προς την αγορά χονδρικής ε, και πλέον ήρθαν και ο Lord Mog και η Τζέν. Ε, με χαρά λοιπόν θα τους δώσω το λόγο προκειμένου να σας παρουσιάσουν το κλάδο της μελέτης μας που αφορούσε την προστασία των καταναλωτών και την ενίσχυση των καταναλωτών. Σας ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση αυτή. Λοιπόν, θα είμαι πολύ σύντομος. Θα αναφερθώ στο δεύτερο τμήμα της παρουσίασης αυτής. Σε αυτή την επόμενη διαφάνεια θα δείτε κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με την όλο και μεγαλύτερη χρήση των εργαλείων σύγκριση, Εργαλεία με τα οποία τελικά κερδίζουμε όλο και περισσότερου ε, πελάτε, καταναλωτέ, ασχολούνται και ενδιαφέρονται για αυτή την όλη διαδικασία. Είναι αρκετά αργή όμω η διείσδυση των εργαλείων αυτών σύγκριση, και πολλέ φορέ οι πληροφορίε που δίνονται βλέπουμε ότι είναι ακριβεί και ότι όντω οι καταναλωτέ μπορούν και κάνουν αξιόπιστε συγκρίσει. Η γενικότερη εντύπωση και μάλιστα ήμουν τώρα σε μια διάσκεψη που οργάνωσε η για τα καταναλωτικά ζητήματα και βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλοί καταναλωτέ ακόμα οι οποίοι λαμβάνουν λογαριασμού που φέρουν πολύ πολύπλοκε τελικά πληροφορίε. Δεν καταφέρουν να επικεντρωθούν αμέσω λοιπόν στα πιο σημαντικά ζητήματα του λογαριασμού του. Το έθιξα το ζήτημα αυτό γιατί τι ε, προηγούμενε εβδομάδε είδα ότι ε, καθότι λαμβάνουμε όλο και περισσότερο συνδυασμένα προϊόντα. Επιχειρήσεις δεν προσφέρουν πλέον μόνο ενεργειακά προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και τηλεπικοινωνιακά προϊόντα και το καθεξής. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όσο περισσότερο είναι συνδυασμένο το προϊόν το οποίο παρέχεται, τόσο πιο δύσκολη είναι και η σύγκριση των λογαριασμών ενέργειας, ιδίως όσον αφορά την συνιστόσα, το τμήμα που αναφέρεται καθαρά σε ενεργειακά ζητήματα και ενεργειακές υπηρεσίες. Γιατί βλέπετε τελικά ότι πολλές φορές τα πράγματα είναι αρκετά πολύπλοκα και θα πρέπει να μπορούμε να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Για ποιο λόγο τώρα υπάρχει τόσο μεγάλη απόκληση και διαφορά από τη μία, άλλη, από τη μία χώρα στην άλλη όσον αφορά την πρόοδο που είχε σημειωθεί στο ζήτημα αυτό της διαφάνειας και της ενημέρωσης. Οι πληροφορίες που δίνονται μέσω των εφιών μετρητών είναι πληροφορίες χρήσιμες, αξιόπιστες. Ε, οι συσκευές αυτές μπορούν να προσαρμοστούν επίσης ε, στην εξέλιξη της παροχής ενέργειας. Ξέρετε ότι ε, σε πολλά κρατημέλη ενδιαφερόμαστε βέβαια και για τους λεγόμενους ευάλωτους καταναλωτές στις σκανδιναβικές χώρες, στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Μπορεί η παροχή ενέργειας αυτούς να περνάει και από τα συστήματα κοινωνικής ασφάλειας αλλά ξέρετε ότι πολύ συχνά οι ρυθμιστικές αρχές στον τομέα της ενέργειας καλούνται να κάνουν και κάτι ακόμα, να προστατεύσουν τους λεγόμενους ευάλωτους καταναλωτές. Και την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον το ζήτημα αυτό έχει γίνει πολύ σημαντικό για διάφορες χώρες και μας έχει απασχολήσει. Βλέπετε στοιχεία σε αυτή τη διαφάνεια. Βλέπετε εδώ πέρα ποιοι είναι εκτεθειμένοι, όχι αναγκαστικά μόνο ηλικιωμένοι, τα άτομα αναπηρίε, τα άτομα με εξαρτώμενα μέλη, με παιδιά κτλ. Το ζήτημα λοιπόν αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν έχει να κάνει καθαρά και μόνο με το ζήτημα της ενέργειας. Αυτά είχα να πω κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε, ο κύριος Μπλέινι. Να προσθέσω κι εγώ κάτι ακόμα ως ρυθμιστικές αρχές όλο και περισσότερο θα πρέπει να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε την όλο και πιο πολύπλοκη κατάσταση προκύπτει για τους καταναλωτές. Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν κεντρικό πλέον ρόλο. Έχουμε όλο και πιο νέες τεχνολογίες που φτάνουν, έχουμε το διαδίκτυο των πραγμάτων, πολλές άλλες τεχνολογικές εξελίξεις και όπως είπε και ο Τζον είναι πάρα πολύ σημαντικό να αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε και με άλλες ρυθμιστικές αρχές όπως για παράδειγμα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών καθώς επίσης και με τους υπόλοιπους οργανισμούς και υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να καταφέρουμε να κρατήσουμε όντως ως βασικό μας μέλημα τον καταναλωτή και να καταφέρουμε να ανακτήσουμε τελικά την εμπιστοσύνη του. Θεωρώ ότι ε, η εργασία που έχει κάνει ο Τζον είναι εξαιρετική και πραγματικά θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για όλη αυτή τη σκληρή σου εργασία ιδίω για την εργασία που έκανε επικεντρώμενο στου καταναλωτέ. Και θα προσπαθήσω και εγώ με τη σειρά μου σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει το πολύ θετικό σου έργο. Ευχαριστούμε πολύ. Όντως δεν συμβαίνει πολύ συχνά να έχουμε έναν διάδοχο τελικά ο οποίος επενεί τόσο πολύ τον προκάτοχό του. Πολύ ωραία λοιπόν. Έχουμε τον απερχόμενο πρόεδρο του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας. Έχουμε επίσης και τον νέο πρόεδρο. Να λοιπόν, χρυσή ευκαιρία, κυρίες και κύριοι, να θέσετε ερωτήσεις. Ποιος θέλει να ξεκινήσει πρώτος. κύριος Πόχε και ο κύριος Κόλιτσεκ στη συνέχεια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με ιδιαίτερη χαρά σας ξαναβλέπω κύριε Διευθυντά και θα ήθελα ειλικρινά να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση που κάνετε όσον αφορά την ετήσια αυτή έκθεση παρακολούθησης του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας. Προφανώς υπάρχει ακόμα ένα περιθώριο βελτίωσης. Τρία πράγματα μπορούμε να αντλήσουμε ως διδάγματα από την έκθεση. Πρώτον, οι λεγόμενοι ευφυείς μετρητές δεν χρησιμοποιούνται επαρκώ. Ένα 25% μόνο των οικοκυριών χρησιμοποιεί αυτού του μετρητέ. Και ωστόσο, βλέπουμε ότι θα μπορούσαν να δώσουν πολύ χρήσιμε πληροφορίε στον καταναλωτή όσον αφορά το κόστο τη ε, κατανάλωση ενέργεια. Και κάτι ακόμα το οποίο προκύπτει από την έκθεση αυτή είναι ότι δεν έχουμε ακόμα επαρκή εργαλεία για την παροχή διαφανών πληροφοριών προς τον καταναλωτή, ο οποίος να μπορεί έπειτα να προχωρεί και σε αξιόπιστες συγκρίσεις. Από την ε, μελέτη άλλωστε προκύπτει ότι στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας υπάρχουν 10 διαφορετικές ε, ε, πληροφορίες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο μάλιστα είναι 14 πληροφορίες που είναι άσχετες ή ακατανόητες. Δυσδιάκριτο το τι ακριβώς ε, σημαίνουν όλες αυτές τις πληροφορίες. Γι' αυτό και χρειάζεται επιτέλους να ενισχύσουμε τη διαφάνεια στον τομέα και νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει επιτέλους να επιληθεί στο, στο πλαίσιο της οδηγίας για την εσωτερική, αγορά. Ε, νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να θεσπιστούν το συντομότερο δυνατό ε, μέτρα για τη βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών. A v té zprávě se vyskytují velmi zajímavá data na straně 6. Ευχαριστώ. Για την ε, σελίδα 6 της μελέτης σας θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Κύριε Χειρογλυκά. Τα σλοβενικά τα μιλάω λιγάκι, δεν μπορώ να... Τώρα, αν προτιμάτε Γαλλικά, ε, γαλλικά θα μπορούσα να συνεχίσω, αν θα μπορούσα να συνεχίσω και ισπανικά. Στη σελίδα 6 βλέπουμε το benchmark capacity, την, το δυναμικό αναφοράς ε, για την υψηλή τάση και τη μεταφορά ενέργειας. Εκεί υπάρχουν ε, διασυνδέσεις μεταξύ Πολωνίας, Τσεχίας, Γερμανίας, Πολωνίας, Σλοβακίας, Πολωνίας, Πολωνίας, Βαλτικών χωρών. Είναι πολύ ενδιαφέρον Αυτές οι διασυνδέσεις μέσω της Πολωνίας ε, συχνά μένουν αχρησιμοποιητές. Ακριβώς αυτό είπατε κι εσείς. Ή ο διαδοχός σας. Γιατί συμβαίνει αυτό. Το ξέρω, το συζητούσαμε τις, με τους διαχειριστές μας στην Τσεχία. Έχω ένα ερώτημα λοιπόν για αυτό το θέμα. Θα ήθελα να ακούσω λοιπόν την απάντησή σας. Γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί μιλάτε συνεχώς για την αγορά. Και εδώ είναι το σύνορο, το οποίο προφανώς είναι αδιάβλητο. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Αυτά τα τερματική Οι αυτοί τερματικοί σταθμοί που χτίζονται εξοδεύοντας τεράστια ποσά με την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών Ταμείων Μιλάμε για τερματικούς σταθμούς ε, υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Πώς επηρεάζουν αυτοί οι τερματικοί σταθμοί την αγορά του φυσικού αερίου, την, τον, την παροχή και τις τιμές του φυσικού αερίου. Ξέρω και την απάντηση μάλιστα. Θα ήθελα να την ακούσω όμως από εσά. Ευχαριστώ. Wow, πολλές γλωσσικές ικανότητες έχετε. Μας εντυπωσιάζετε. Ε, δεν ξέρω αν ο επόμενο ομιλητή μπορεί να είναι στο ίδιο επίπεδο γλωσσικών ικανοτήτων. Δεν θα προσπαθήσω καν, λέει ο κ. Πίτερσεν. Καταρχά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Ποτότσνικ και τον ε, Λόρδο Μόγ για την θαυμάσια συνεργασία τα τελευταία δύο-τρία χρόνια. Πολύ χρήσιμο να ακούμε πάντα τις σκέψεις σας και τις απόψεις σας για αυτό το πολύ κρίσιμο σημείο. Σας ευχαριστώ λοιπόν και τους δύο για το θέμα αυτό. Φαντάζομαι και με τον ε, διάδοχό θα συνεργαστούμε πολύ καλά. Πάμε στη σελίδα 6 της παρουσίασής σας για την, την αναλογία ανάμεσα στο διασυνοριακό δυναμικό και στο δυναμικό αναφοράς. Με εντυπωσιάζουν αυτά τα νούμερα. Από ό,τι θυμάμαι, Αλμπέρτο, είπες ότι ο μέσος όρος Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι περίπου το 50%. Ο λόγος δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε μόνο το μισό δυναμικό που έχουμε. Αυτό είναι ένα απλό ζήτημα, αλλά το υποτιμούμε, υποτιμούμε τη σημασία του. Εξού και η ερώτησή μου προς εσάς. Αν θέλουμε να ποσοτικοποιήσουμε τα ωφέλη από το να φτάσουμε από το 50% όχι στο 100% αλλά τουλάχιστον να πάμε από το 50% σε κάτι παραπάνω που να είναι ρεαλιστικό. Και δεν θα φτάσουμε από τη μια μέρα στην άλλη, ας πούμε, σε αυτά τα επίπεδα, έτσι, ούτε καν σε ένα χρόνο. Αλλά είναι πάντως ένας τομέας που θα έπρεπε να κάνουμε κάτι για τον Ευρωπαίο καταναλωτή και Ευρωπαίο πολίτη, μέσω της κατάλληλης νομοθεσίας που θα εξασφαλίζει την ελεύθερη ροή ενέργειας. Οποτεδήποτε συζητάμε ε, τα ωφέλη της ενιαίας αγοράς στο Κοινοβούλιο, ειδού η απόδειξη ότι δεν έχουμε φτάσει σε καμία περίπτωση εκεί που θα έπρεπε. Είμαστε στο 50%. Και στη δεξιά στήλη βλέπω κάποια νούμερα, τα οποία είναι ακόμα πιο ανησυχητικά. Πιο χαμηλά από το 50%. Έχετε ποσοτικοποιήσει πιθανά ωφέλη από το να αυξηθεί ο λόγος αυτός. Θεωρητικά, τι θα μπορούσαμε να δώσουμε στους Ευρωπαίους εάν είχαμε τη σωστή νομοθεσία και την εφαρμόζαμε. Ευχαριστούμε κύριε Πίτερσεν. Και τώρα κάποια σχόλια ή μάλλον κάποια, θα ακούσουμε και λίγα βαβαρικά από την κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ. Δεν θα μιλήσω βαβαρικά, θα μιλήσω την ε, ε κοινή γερμανική. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω ε, για την παρουσίασή σας και για την ε, πολύ συχνή ανταλλαγή απόψεων που έχουμε εδώ στην Επιτροπή μας μαζί σας. Δύο ερωτήματα. Πρώτον, πόσο είναι η, πώς είναι η προθυμία αλλαγής παρόχου μεταξύ των καταναλωτών. Αναφερθήκατε σε ένα ποσοστό 20% αλλά ε, πόσο, πόσο είναι το ποσοστό αυτό στα επιμέρους κράτους, κράτη-μέλη. Πόσο, πώς είναι η προθυμία των, των ίδιων των καταναλωτών να αλλάζουν παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Έχετε σχετικά στοιχεία και δεύτερον. Γνωρίζετε ότι συζητούμε αυτό το διάστημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το πακέτο για την καθαρή, καθαρή ενέργεια. Πολύ πρόσφατα λοιπόν ε, εγκρίναμε και την πρόταση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ένα ακαθόδες θέμα. Εσείς ε, έχετε στοιχεία για το ποιε είναι οι επιπτώσεις των ε, ενισχύσεων για τις ανανεώσιμες πηγέ ανέργεια ε, στις τιμές τη ηλεκτρική ανέργειας στη Γερμανία. Ε, έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια επιδοτήσεις ύψους έως και 20 δισεκατομμυρίων κατέτος για τις ανανεώσιμες πηγές ανέργειας. Έχετε λοιπόν εσείς στοιχεία για το ποιες είναι οι επιπτώσεις της ε, ε, ανάπτυξης και της υποστήριξης των ανανεώσιμων πηγών, πηγών ενέργειας στις τιμές ε, που πληρώνουν οι καταναλωτές στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να θέσω δύο ερωτήματα. από το, στο, προς τον κύριο Ποτότσνικ, ε, αντίστοιχη με τη κυρία Νίπλερ, οι Γερμανοί καταναλωτές πληρώνουν τη δεύτερη ψηλότερη τιμή για την ηλεκτρική ενέργεια, το ηλεκτρικό ρεύμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε κάποια ιδέα ε, του ποσοστού στο οποίο οφείλεται στην έλλειψη ανταγωνισμού του ποσοστού της τιμής. Και μια δεύτερη πιο φιλοσοφική ερώτηση προς τον Λόρδο Μόγκ, ο οποίος εντάξει, έχει εμπειρία για να απαντήσει αυτή τη δύσκολη ερώτηση. Μια και φεύγεται ίσως θα μπορούσε να μου απαντήσει ειλικρινά. Θα βρείτε το κουράγιο. Το ερώτημα είναι, μιλάμε πάντα για την, για την Ενεργειακή Ένωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. προσπαθούμε να κάνουμε εκεί πέρα ό,τι κάναμε και στην ε, ενιαία αγορά. Από την άλλη λέμε ότι κάθε χώρα καθορίζει το ενεργειακό της μείγμα. Εξού και η ερώτησή μου τώρα. Θα είμαστε σε θέση ποτέ να φτάσουμε σε μια πραγματική ενεργειακή ένωση αφήνοντας ε, μια κυβέρνηση της, και όχι την αγορά, μια κυβέρνηση ενός κράτους μέλους να αποφασίσει για το ενεργειακό μείγμα. Μπορεί να γίνει αυτό πράγμα. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Θα απαντήσω σε εκείνες που συνδέονται με την αγορά τη χοντρική. Ο κύριος Κούλιτσεκ. Γιατί έχουμε χαμηλά επίπεδα δυναμικού, διαθέσιμου δυναμικού. Και ο κύριος Πέτερσεν νομίζω αναφέρθηκε σε αυτό αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εγγενής ε, διακριτική μεταχείριση εις βάρος των διασυνοριακών ροών υπέρ των εσωτερικών ροών. Αυτό έχει να κάνει το σχεδιασμό της αγοράς. Οι εσωτερικές ροές, εντός δηλαδή, μίας ζώνης υποβολή προσφορών δεν, δεν αντιμετωπίζουν περιορισμούς. Κάθε ζώνη που προσδιορίζεται στην πραγματικότητα υποστηρίζεται και από του ε, TSO. Όταν κοιτάμε τις διασυνοριακές ε, ροές, έχουμε, όταν έχουμε ε, σύνορο εκεί, στις, τα bidding zones, ε, εκεί έχουμε πρόβλημα. Αν το σύστημα σε μία bidding zone δεν είναι σε θέση να υποστηρίξει το επίπεδο ροών που καθορίζονται, σε κάθε, τότε, σε, τότε το, η ροή χρησιμοποιεί άλλα μονοπάτια και συμπληρώνει το δυναμικό στα άλλα μονοπάτια. Δηλαδή, αυτό το δυναμικό δεν μπορεί να δοθεί για εμπόριο, γιατί απορροφάται από ροές που δεν απορρέουν από το εμπόριο ανάμεσα σε αυτά τα σύνορα, αλλά σε άλλα σύνορα ή εντός κάποια συγκεκριμένης ε, ζώνης υποβολής προσφορών. Χρησιμοποιείται λοιπόν το δυναμικό, αλλά όχι για το εμπόριο, αλλά για να υποστηρίξουμε άλλες ροές τα loop flows όπως τα λέμε. Και δεν υπάρχουν λοιπόν, δεν μπαίνουν αυτές οι ροές προς εμπορία. Ελπίζω να είναι χρήσιμη η απάντηση. Αυτό που έχουμε στη σύστασή μας, προσπαθούμε να αποφύγουμε αυτές τις διακρίσεις. Δηλαδή το δυναμικό το οποίο υπάρχει για το διασυνοριακό εμπόριο να υπολογίζεται ως απομεινάρι αυτή τη στιγμή οι εσωτερικές ανταλλαγές έχουν καλυφθεί. Θέλουμε τα διασυνοριακέ και εσωτερικές ροές να τις έχουμε στο ίδιο επίπεδο. Και θα πρέπει να λάβουμε μέτρα και στις δύο περιπτώσεις εάν ξεπεράσουμε το δυναμικό του δικτύου. Αλλά τουλάχιστον να μην υπάρχουν ίδιες διακρίσεις. Και τη τρίτη αρχή που δεν έχει ακόμα ενσωματωθεί στην νομοθετική πρόταση είναι το ποιος θα πληρώσει για αυτές τις δράσεις βελτίωσης ή διόρθωσης. Αν η χρήση ή η ζήτηση α, του δικτύου ξεπερνάει το δυναμικό. Υγροποιημένο φυσικό αέριο και τα τερματικά του. Μπορώ να σας πω πολλά, να σας δώσω ένα παράδειγμα και φαντάζομαι τα ξέρετε όλα αυτά, μια και ξέρετε την απάντηση, αλλά σας δώσω και εγώ την απάντηση. Όταν η Λιθουανία ανέπτυξε το δικό της θερματικό. Πριν φτάσει το πρώτο φορτίο φυσικού αερίου, η τιμή του εισαγόμενου φυσικού αερίου με το πρώτο φορτίο μειώθηκε θεαματικά. Για μένα αυτό είναι η απόδειξη του ανταγωνισμού. Και επίση ε, αντιμετωπίστε και το πρόβλημα ασφάλεια ε, ανεφοδιασμού. Ε, υπάρχουν περισσότεροι δρόμοι για το φυσικό αέριο για να έρθει έρχεται το φυσικό αέριο στην Ευρώπη από διαφορετικές πηγές και φυσικά δημιουργεί ανταγωνιστική πίεση στις καλά εγκατεστημένες πηγές και πιέζει αυτές τις καλά εγκατεστημένες πηγές παροχής αερίου. Κύριε Χέγκλ και κύριε Πέτερσεν, δεν μπορώ να σας δώσω εκτίμηση του πόσο το, το, τμήμα, του τμήματος της τιμής οφείλεται στο σχεδιασμό της αγοράς ή ποιο θα ήταν το όφελος από το να εξαλείψουμε κάποια από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Το, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι με τη διασύνδεση για να φτάσουμε εδώ που είμαστε τώρα δηλαδή, εκτιμούμε ότι δίνουμε ένα δισεκατομμύριο το χρόνο στους Ευρωπαίους καταναλωτές. Αν το διαιρέσετε με όλο το λογαριασμό που πληρώνουμε για το φυσικό εμπόριο είναι 0,000%. Παρ' όλα αυτά είναι ένα ε, δισεκατομμύριο. Δεν φτιάξαμε καινούριε γραμμέ διασύνδεση, δεν βάλαμε γραμμέ, α πούμε, από ατσάλι ή χαλκό ή οτιδήποτε. Απλώ βελτιώσαμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε αυτό που έχουμε ήδη. Δεν το χρησιμοποιούμε στο 100% αυτού που θα μπορούσε μηδενικά, αλλά λειτουργεί καλύτερα η αγορά. Υπολογίζουμε ότι 220, 250, 280 εκατομμύρια ευρώ μπορούμε να κερδίσουμε αν ε, επεκτείνουμε τις διασυνδέσεις των αγορών στα υπόλοιπα σύνορα που δεν είναι διασυνδεδεμένα. Περί αυτού πρόκειται λοιπόν. Μιλάμε για εκατομ... εκατοντάδες εκατομμύρια, ίσως και δισεκατομμύρια. Εάν ε, λάβουμε υπόψη μας και το δυναμικό που έχουμε. Ορισμένες χώρες όμως τότε μπορεί να αλλάξουν το μείγμα, ή μάλλον ε, το σχεδιασμό της αγοράς για να υπάρχει μεγαλύτερη υποδοτικότητα. Αυτό θα το αποφασίσουν οι χώρες όμως. Τέλος. Κυρία Νίμπλερ. Ποια είναι η επίπτωση των ανεώσιμων πηγών ενέργειας στις ε, τιμές χοντρικής με περισσότερες ανανεώσιμες, ε, οι νέες ανανεώσιμες πηγές είναι ποικίλε και επομένως θα αυξηθεί η ποικιλομορφία της αγοράς χοντρικής. Αυτό δημιουργεί μια πρόκληση, ένα πρόβλημα, γιατί χρειαζόμαστε μια πιο ευέλικτη αγορά χοντρικής. Από την άλλη, μπορεί να έχουμε πιο ασταθείς τιμές, γιατί όταν φυσάει ο άνεμος, ας πούμε, θα έχουμε ενέργεια από τις ανανεώσιμες αυτές. Όταν δεν υπάρχει άνεμος θα πρέπει να αναζητήσουμε άλλες ανανεώσιμες για να καλύψουμε αυτό το, αυτή την ανάγκη και μπορεί να αυξηθεί το κόστος. Μετά από πολλά χρόνια όπου δεν υπήρχαν ε, κορυφώσεις τιμών, πέρυσι είχαμε αυξήσει των τιμών. Οφείλεται και σε άλλα πράγματα ίσω, αλλά στο μέλλον θα έχουμε πιο ασταθεί τιμέ μέχρι να φτάσουμε σε κάποιο επίπεδο όπου το σύστημα θα εξυπηρετείται μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια και τότε θα δούμε με τι θα μοιάζουν οι τιμέ. Αλλά αυτό δεν θα γίνει πριν από 15 με 20 χρόνια. Οπότε έχουμε χρόνια να το σκεφτούμε. Και πριν δώσω το λόγο στο Λόρδο Μόγκ, είναι η τελευταία έκθεση παρακολούθησης αυτή που, παρακολου... παρα... παρουσίασα, γιατί μέχρι του χρόνο θα έχω τελειώσει τη θητεία μου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξη προς το πρόσωπό σας και προς τον οργανισμό μου αυτά τα 7-7,5 χρόνια. Νομίζω ότι σιγά σιγά περνάμε σε μία άλλη εποχή σε σχέση με αυτά που είπε ο Αλμπέρτο και απαντώντας τον κύριο Πέτερσεν ποια είναι η σχέση μεταξύ της κοινότητας των ρυθμιστών του οργανισμού μας όλα αυτά τα χρόνια και προτού καν δημιουργηθεί ο οργανισμός μας αυτός. Πρέπει να σας πω ότι μεταξύ μόνο συνεργασία ήταν πάρα πολύ υποφελής για τον οργανισμό, για τις ρυθμιστικές αρχές και ανέκαθεν είχαμε και την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πάντα σας έλεγα ότι είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Να και εγώ με τη σειρά μου σε κάποια επιμέρους σημεία. Όσον αφορά τους ευφύης μετρητές, πρέπει να σας πω ότι παραλύω κάπως από την πολυπλοκότητα του συστήματος και από τη σχετική νομοθεσία. Ξέρετε ότι η ανάλυση κόστους ωφέλους πρέπει πάντα να είναι θετική και δεν είναι πάντα θετική. Αν έχουμε μία ευρία επέκταση των εφιών αυτών μετρητών σε πάρα πολλές χώρες, μπορεί να οδηγηθούμε απότομα σε πολύ υψηλέ δαπάνες και ενδεχομένω το σύστημα πολύ γρήγορα να καταστεί παροχημένο εξαιτία των τεχνολογικών εξελίξεων. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα σύστημα ιδιαίτερα πολύτιμο για τι ίδιε τι εταιρείες παροχής ενέργειας, καθότι συλλέγουν κατά αυτόν τον τρόπο δεδομένα πολύ πιο γρήγορα και χωρί να χρειάζεται καν να πάνε στα σπίτια των καταναλωτών. Για τους μεμονωμένου τώρα καταναλωτέ, πάλι διστάζω να το πω εν μέρη, γιατί από προσωπική πλευρά. Αυτή τη στιγμή αρχίζει κανείς να βλέπει την κατανάλωσή του, την προσέχει στην αρχή και μετά λίγο την αμελεί. Ένα σύστημα λίγο πιο πολύπλοκο θα καταφέρει τελικά να μας δώσει πιο αξιόπιστες και χρήσιμες πληροφορίες προκειμένου να μπορούμε πραγματικά να ελέγχουμε καλύτερα την κατανάλωσή μας. Στον κύριο Χατσέκ τώρα. Νομίζω ότι η ενημέρωση είναι πάντα πολύ σημαντική σε σχέση με την κατανάλωση που έχει λάβει η χώρα δηλαδή. Νομίζω πάντως ότι μία από τις σημαντικότερες δυσκολίες που συναντάμε ως ρυθμιστικές αρχές και όχι μόνο, είναι το ότι υπάρχουν πάρα πολλές πλέον πληροφορίες, ένας τεράστιος όγκος πληροφοριών και πέρα από αυτό το σημαντικότερο πρόβλημα είναι ότι βρισκόμαστε ακόμα σε ένα αρχικό στάδιο συνδυασμένων προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό θα καταστήσει την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη απευθυνόμενος και στον πρώην πρόεδρο της Επιτροπής ΙΤΡΕ, ε, να τον ευχαριστήσω καταρχάς για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε στο παρελθόν. Όσον αφορά τα δεδομένα, έχουμε μια σειρά από δεδομένα για την κατανάλωση των οικοκυριών και βλέπουμε εδώ πέρα ότι είχαμε μια αύξηση από το 5% το 2011 σε 6,4%. Αυτά τα δεδομένα έχουν να κάνουν με την αλλαγή που κάνουν οι καρτιναλωτέ όσον αφορά το ενεργειακό του μείγμα. Βλέπετε λοιπόν το ποσοστό ακόμα παραμένει πολύ χαμηλό. Αυτό το πρόβλημα ήταν σημαντικό, δυσεπίλητο στην αρχή και εμεί ω ρυθμιστικέ αρχές προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Βλέπουμε ότι η αλλαγή του παρόχου έχει οδηγήσει τις ρυθμιστικές αρχές να κάνουν τις απαραίτητες προσαρμογές και αυτές για να μπορούν να παρακολουθούν καλύτερα την εξέλιξη των τιμών. Σε ορισμένες χώρες έχουμε ήδη συγκρίσιμα δεδομένα αξιόπιστα τα οποία χρησιμοποιούμε και βάσει των οποίων μπορούμε να πούμε ότι αξίζει κανείς να αλλάξει πάροχο, αλλά αλλού πάλι τα στοιχεία είναι λίγο πιο προβληματικά και κάπως ανεπαρκή. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν κύριε Διευθυντά, κύριε Πρόεδρε. Αυτή είναι η τελική σας, τελευταία σας μάλλον συνεδρίαση εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να πω κάτι για το ενεργειακό μείγμα πρωτού ολοκληρώσω. Πρέπει να σας πω ότι όσον αφορά την ιστορική αγορά, λυπάμαι πάρα πολύ για το Brexit. Αρχίσουμε αυτή τη στιγμή να βλέπουμε ποια, θα είναι η κατάσταση μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ουσιαστικά όλα τα δεδομένα δείχνουν ε, ότι σε όλο αυτό το φάσμα από την εσωτερική αγορά στην Ενεργειακή Ένωση η ολοκλήρωση τελικά είναι αυτή που καθιστά τις αγορές πολύ πιο αποδοτικές και πιο επωφελείς τελικά για τους καταναλωτές. Δεν ξέρω γιατί αύξηση θα μιλήσουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένα 4% ενδεχομένω. Όλα τα επιχειρήματα συγκλίνουν στο ότι η ολοκλήρωση προφανώς, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και η ολοκλήρωση των αγορών ενέργειας είναι προς το όφελος των κρατών και των καταναλωτών. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει και απαραίτητη πολιτική βούληση και δυστυχώ υπάρχουν πολλέ κυβερνήσει οι οποίε δεν θέλουν να εγκαταλείψουν την κυριαρχία του σε έναν τομέα όπω όπως η ενέργεια. Για παράδειγμα, στην Γαλλία ένα μεγάλο μέρο τη ηλεκτρική ενέργεια απορρέει από την πυρηνική ενέργεια. Αυτός είναι ένας λόγος που ορισμένες χώρες δεν θέλουν να κάνουν εκχωρήσεις στον τομέα της ενεργειακής τους κυριαρχίας. Πάντως, ε, προϊόντος του χρόνου και όσο θα ολοκληρώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι όλο και περισσότερες χώρες θα συνειδητοποιήσουν τα ωφέλη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στον τομέα της ενέργειας. Νομίζω ότι αυτό θα επικρατήσει στο τέλος. Πόσο θα χρειαστεί βέβαια για να φτάσουμε στο σημείο αυτό. Πόσα χρόνια θα χρειαστούν προκειμένου να υπάρχει ένας, μια ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή. Νομίζω ότι μιλάμε για διψήφιο αριθμό. Ενδεχομένως σε 15-20 χρόνια. Και είδατε ότι ουσιαστικά αναφέρομαι σε μια περίοδο όπου ενδεχομένω να μην με κάνει ζωή. Μα μην, μην είστε τόσο απεσιόδοξο, λέει ο πρόεδρο. Καταρχά, Νορδεμόγκ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική σας αυτή παρέμβαση. Όντως, συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά στο παρελθόν με τον οργανισμό σας. Μας έχετε δώσει εξαιρετικές συμβουλές και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εσάς, κύριε Ποτότσνικ, για την τελευταία αυτή παρουσίασή σας στην, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε σχέση με την εργασία που κάνει ο συγητή μα ο κύριο Πέτερσεν στα πλαίσια του, της Επιτροπής μας και να ευχηθώ καλή τύχη και κάθε επιτυχία στον κύριο Μπλέινι και θα έχετε συνειδητοποιήσει βέβαια ότι έχουμε εμεί πολύ υψηλέ προσδοκίε από εσά σε σχέση με τα θετικά βέβαια που είπατε και για τον προκάτοχό σα. Είμαστε ακόμα πιο απαιτητικοί. Κυρίε και κύριοι, περάσουμε τώρα σε ένα παρεμφερέ ζήτημα Ας περάσουμε σε ένα παρεμφερές ζήτημα. Πάλι θα μιλήσουμε για τον Νέισερ. Ξέρετε ότι υπήρξε μια αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου Μάσα. Ο κύριος Πόχε και Πέτρεσεν ήταν μέλη τη αντιπροσωπείας αυτής, οι οποίοι θα μας κάνουν μια σύντομη παρουσίαση των απορισμάτων τους. Κύριε Πέτρεσεν, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ξέρετε ότι σας έχω δώσει και ένα έγγραφο ενημερωτικό, ελπίζω το έχουν λάβει τα μέλη της Επιτροπής μας. Οι πληροφορίες είναι τόσες, τόσο πολύτιμες στο έγγραφο αυτό και πραγματικά σας επιτρέπει να έχετε μια πιο σφαιρική εικόνα των δραστηριοτήτων που, στις οποίες προχωρήσαμε και όλων αυτών των εκδηλώσεων στις οποίες συμμετείχαμε. Πάντα είναι μεγάλη χαρά να επισκεπτόμαστε τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας το προσωπικό είναι ιδιαίτερα καταρτισμένο και θα έλεγα κύριε Πρόεδρε και νομίζω ότι μπορώ να το πω παρουσία του κυρίου Ποτότσνικ, ο οποίο δίνει τώρα στο Προεδρείο, ότι ήταν πραγματικά προνόμιο για μας, τιμή για μας, να μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με ένα τόσο προσιλωμένο, πρικισμένο τελικά προσωπικό, το οποίο πραγματικά συνεργάζεται με τους νομοθέτες εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήταν πραγματική ευχαρίστηση για μας. Στα πλαίσια λοιπόν του εγγράφου αυτού που σα έχουμε διανύμει, βλέπετε τα πιο σημαντικά σημεία τα οποία θίξαμε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας και τα οποία θα μας απασχολήσουν βέβαια και στο μέλλον. Σας καλώ λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι να διαβάσετε το έγγραφο αυτό γιατί πραγματικά θα σας δώσει μια πολύ καλή γενική επισκόπηση των σημαντικότερων ζητημάτων της συνεργασίας μας με τον Acer. Πέρα από όλα αυτά μας δόθηκε επίσης και η δυνατότητα να συναντήσουμε το προσωπικό του οργανισμού και είχαμε μάλιστα και τη δυνατότητα να απαντήσουμε σε ερωτήσεις του προσωπικού ή να τους υποβάλουμε και εμείς ερωτήσεις. Αυτό ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον, ιδιαίτερα χρήσιμο πάλι για μας. Μπορέσαμε κατά αυτόν τον τρόπο να συναντήσουμε πολλά μέλη του προσωπικού, του οργανισμού και είδαμε πραγματικά πόσο επαγγελματικά και με την συνειδησία επιτελούν το, καθέ, το καθήκον τους. Και για τη δυνατότητα αυτή λοιπόν σας ευχαριστώ πολύ. Είναι σαφές ότι για μία ακόμα φορά αυτό που μας απασχόλησε ήταν ο προπολογισμό, η οικονομική κατάσταση του οργανισμού, έχοντας δει πώς εργάζονται οι άνθρωποι σε αυτόν τον οργανισμό και πόσο σημαντικά είναι τα καθήκοντά τους. Το να έχει κανείς λοιπόν τη δυνατότητα να πηγαίνει και να επισκέπτεται προσωπικά τον οργανισμό δημιουργεί πολύ έντονες εντυπώσεις. Και θα ήθελα πραγματικά να διαβιβάσω εδώ πέρα προς συναδέλφους μου πόσο επίγει τελικά πόσο επίγει να δώσουμε τους απαραίτητους πόρους στον οργανισμό αυτό, δεδομένων των τιτάνων καθηκόντων που καλούνται να επιτελέσουν. Ξέρετε ότι μιλούσαμε μόλις τώρα για τη σημαντική τη σημασία της ολοκλήρωσης των ενεργειακών αγορών. Αυτό είναι ένα πράγμα. Αυτή τη στιγμή οι αγορές ενσωματωθούν και ολοκληρωθούν. Πρέπει να υπάρχει και ένας οργανισμός ο οποίος να επιβλέπει, να επιτηρεί όλες αυτές τις δραστηριότητες στον τομέα της ενέργειας. Ε, αυτό ακριβώς κάνει ο Acer και προφανώς χρειάζεται τους απαραίτητους πόρους για να επιτελέσει το έργο του. Είναι σημαντικό να το γνωρίζουν αυτό οι συνάδελφοι στην Επιτροπή μας. Όλα αυτά για να σας πω λοιπόν κύριε Πρόεδρε ότι ήταν τεράστια ευχαρίστηση για μένα να επισκεφθώ τον Acer, τον οργανισμό αυτό στην πανέμορφη Λιουμπλιάνα και θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω και τον Διευθυντή και το προσωπικό του οργανισμού αυτού για τις επαφές που είχαμε και για άλλη μια φορά καλό τους συναδέλφους να διαβάσουν το πολύ καλό αυτό έγγραφο που έχουμε συντάξει και το οποίο ενημερώνει για τις δραστηριότητές μας εκεί. Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλα σχόλια από τους συναδέλφους για το θέμα αυτό. Δεν φαίνεται να υπάρχουν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πέτερσεν. Ο κύριος Πόχε δεν είναι εδώ πια, αλλά φαντάζομαι ότι αυτά που είπατε ε, απηχούν και τις δικές του απόψεις και αυτό που θα ήθελα να κρατήσουμε από σήμερα είναι τα καλά λόγια που ε, απευθύνθηκαν ε, στον κύριο Ποτόστινγκ να μην δράσουν αποτρεπτικά για να συνεχίσει το καλό του έργο. Κάποιες φορές συμβαίνει γι' αυτό. Εν πάση Περνάμε στο επόμενο θέμα, ελεύθερη ροή δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως γνωρίζετε, το Σεπτέμβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια πρόταση κανονισμού για την εξασφάλιση της ελεύθερη ροή δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, πρόσωπο που έχει απασχοληθεί όλη τη ζωή σε αυτόν τον κλάδο, γνωρίζω και βεβαιώνω ότι η ροή δεδομένων αποτελεί τον πυρήνα, την καρδιά της καινοτομίας και της ε, κοινωνίας της πληροφορίας. Στόχος της ε, πρότασης είναι να διευκολυνθεί η διαχείριση, η κυκλοφορία ε, της ροής δεδομένων χωρίς περιορισμού Επί της ουσίας αρμόδια επιτροπή βεβαίως είναι η ΙΜΚΟ, η δική μας επιτροπή γνωμοδοτή και θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Κρασνοντέσκη, τον εισηγητή μας, να παρουσιάσει τα βασικά στοιχεία της γνωμοδότησής του σε πέντε λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε μόλις και εσείς, η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία αποτελεί σημαντικότατο τμήμα και κεφάλαιο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Διότι η ψηφιακή ενιαία αγορά και η σχετική στρατηγική περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία. Ο, βασι... Ο κοινός παρανομαστής όμως είναι τα προσωπικά δεδομένα κάτι που επηρεάζει τη συνολική παραγωγικότητα και αποδοτικότητα της ε, οικονομίας, επηρεάζει την, ε, ε, τους ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕΠ, υπάρχουν μάλιστα ε, επιχειρήσεις μεγάλες, ε, γιγαντιές σε παγκόσμιο επίπεδο που βασίζουν τις ίδιες τους τις οικονομικές δραστηριότητες, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στην ύπαρξη και στην πρόσβασή τους σε προσωπικά δεδομένα. Γι' αυτό και είναι τόσο σημαντικό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκές οικονομίες θα βασίζονται ολοένα και περισσότερο στην ύπαρξη και στην αξιοποίηση δεδομένων και γι' αυτό χαιρετίζουμε θερμότατα την πρόταση αυτή της Κομισιόν καθώς και τα βασικά της στοιχεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά θα έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται και να επεξεργάζονται τα, τους πόρους τους όσον αφορά τα μη προσωπικά ε, δεδομένα ε, βάσει βεβαίως συγκεκριμένων επιχειρηματικών αρχών και αξιών ώστε να μπορούν να προβαίνουν σε σχεδιασμό και χάραξη των επιχειρηματικών τους στρατηγικών. Μέχρι τούδε, όπως γνωρίζουμε όλοι, τα δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα και η σχετική ε, ροή δεν ρυθμιζόταν νομοθετικά. Ε, υπήρχαν λοιπόν διάφοροι περιορισμοί διοικητικού ή άλλου χαρακτήρα που υποχρέωναν ε, τις επιχειρήσεις να αποθηκεύουν δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα σε χώρες όπου έχουν την έδρα τους. Κάτι που αποτελούσε διαχρονικά μεγάλο εμπόδιο όσον αφορά την επιχειρηματικότητα και την ελευθερία του επιχειρήν σε ολόκληρη την ενιαία αγορά. Ενώ αντιθέτως το μόνο, η μόνη κόκκινη γραμμή, ο μόνος περιορισμός θα έπρεπε να είναι η προσωπική ασφάλεια του κάθε Ευρωπαίου πολίτη. Θέλω να πω με άλλα λόγια ότι η συγκεκριμένη πρόταση αποτελεί ένα μόνο από τα βήματα ε, που θα απαιτηθούν προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης ελευθερία ροής δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθώς το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας ε, αφορά μόνο την, ε, την, την, την έδρα. Τα άρθρα 4 και 6 συγκεκριμένα. Ενώ μακροπρόθεσμα η διάταξη αυτή ενδέχεται να αποδειχθεί ε, ανεπαρκής. Γι' αυτό ενδέχεται να χρειαστεί να ανοίξουμε την πρόσβαση ε, και σε βιομηχανικής κλίμακας επεξεργασία δεδομένων. Αν θέλουμε λοιπόν η οδηγία αυτή να επιτύχει πραγματικά τους στόχους της, χρειάζεται να τροποποιηθούν τα άρθρα, το άρθρο 6 κατά κύριο λόγο δεν θα πρέπει να υπάρχουν εμπόδια που θα προκύπτουν από την αυτορύθμιση. Συνεπώ, είναι απαραίτητο να υπάρξει καθοδήγηση και διευθυντήριε γραμμέ όσον αφορά την αυτορύθμιση και θα πρέπει επίση να επισημανθεί ότι η κινητικότητα δεδομένων θα είναι ε, στοιχείο της ε, αρχής ελευθερίας παροχής υπηρεσιών. Να περιλαμβάνονται δηλαδή τα διαλειτουργικά πρωτότυπα, η, αμοιβία, η αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών ποιότητας, ώστε να μην δημιουργηθούν τεχνητά ε, εμπόδια στην ε, κυκλοφορία δεδομένων. Συνοψίζοντας λοιπόν θέλω να πω ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υποστηρίζουμε τη γενική κατεύθυνση της πρότασης της Κομισιόν. Οι δικές μας προσθήκες από εκεί και πέρα θα αφορούν ιδίως την κινητικότητα Και ας ελπίσουμε ο κανονισμός αυτός να τεθεί σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό, ώστε να υλοποιηθεί ε, το συντομότερο δυνατό η συγκεκριμένη ελευθερία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όπως είπα η οικονομική σημασία αυτής της ελευθερίας είναι πάρα πολύ σημαντική ενώ είναι πολύ σημαντική η εν λόγω ελευθερία βεβαίω και για την ολοκλήρωση τη ψηφιακή ενιαία αγορά, όπω είπα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κρασνοντεύσκη για το ΕΛΚ, η κυρία Βυρκούν. Ευχαριστώ. Τρία λεπτά μου δίνετε. Ο χρόνο αγόρευση, Έχω τρία λεπτά. Α, δύο, δύο, μάλιστα. Εντάξει, θα τα πω γρήγορα. Ευχαριστώ τον ε, συντάκτη τη γνωμοδίτησης. Πρέπει να πω ότι δεν έχω πολλά να προσθέσω γιατί συμφωνώ με τα περισσότερα πόσα είπε όσον αφορά το ρόλο των δεδομένων στην ψηφιακή έννοια αγορά γιατί γνωρίζετε ότι πρόκειται μία από τις βασικότερες προτεραιότητες μας να ολοκληρωθεί αυτή η ψηφιακή έννοια αγορά και προφανώς οι ροές δεδομένων αποτελούν βασικό συστατικό ε, της ολοκλήρωσης αυτής της ε, ενιαίας ε, αγοράς. Γνωρίζουμε ότι η ροή δεδομένων βρίσκεται στον πυρήνα ε, των ε, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων και διαφόρων μεγεθών από τον τουρισμό, τη γεωργία, την τεχνολογία πληροφορία και επικοινωνίας καθώς και μια σειρά από άλλους κλάδους. Υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες οικονομικές όσον αφορά την αξιοποίηση των ε, δεδομένων. Πέρσι η αξία της αγοράς δεδομένων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμάται σε περί τα 60 δισεκατομμύρια ευρώ και εκτιμάται επίσης ότι το 2020 η αξία αυτής της αγοράς θα ε, ανέλθει σε, επίπεδα άνω των 100 δισεκατομμύριων ευρώ. Εμπόδια όσον αφορά την ολοκλήρωση της ψηφιακής ψηφιακή αγοράς αγορά είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ε, εμπόδια όσον αφορά την κινητικότητα δεδομένων, τις ε, γεωγραφικούς περιορισμούς για τη χρήση και επεξεργασία δεδομένων που ακόμη υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που δεν συνάδουν με την ιδέα της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Γι' αυτό και πρέπει να αρθούν τα εμπόδια αυτό, αυτά κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ιδίως για τις επιχειρήσεις, καθώς εκείνες είναι αναγκασμένες να διατηρούν έδρα σε διάφορες χώρες, κάτι που είναι πάρα πολύ δαπανηρό. Επίσης, συμφωνώ με το συντάκτη της γνωμοδότησής ότι αυτή η πρόταση είναι ένα πρώτο βήμα, όχι όμως το μοναδικό που απαιτείται προκειμένου να δημιουργηθεί μια πραγματική ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών. Χρειάζονται και άλλα μέτρα προκειμένου να επιτευχθεί η ψηφιακή ενιαία αγορά και στον τομέα της ροής δεδομένων και νομίζω ότι με αφορμή αυτή την πρωτοβουλία θα πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση στο μέλλον για την πρόσβαση στα δεδομένα, την αξιοπιστία, τη φορητότητα των δεδομένων, διότι γνωρίζουμε ότι η ελεύθερη ροή δεδομένων είναι κρίσιμη, ζωτική σημασία για την ψηφιακή μα αγορά. Γι' αυτό και είναι πολύ θετικό το γεγονό ότι έχουμε πλέον δεχτεί αυτή την πρόταση από την Κομισιόν. Ο κύριος Πέτερσεν για τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς χαιρετίζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς ως πολιτική ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια τέτοια πρόταση. Ιδίω όταν βλέπουμε την ανησυχητική αυτή τάση παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου υπάρχουν όλο και περισσότερες απαιτήσει εντοπισμού, εντοπικότητας μάλλον των δεδομένων αυτών. Ξέρετε ότι δεν μπορούν πολλές εταιρείες startup να λειτουργήσουν διασυνοριακά. Ας αποφύγουμε λοιπόν, θα έπρεπε να είχαμε αποφύγει μάλλον αυτόν τον κατακαιρματισμό. Η ελεύθερη ροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι πάρα πολύ σημαντική και για την ασφάλεια. Για παράδειγμα η Εστονία έχει πει ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει μια ψηφιακή πρεσβεία στο Λουξεμβούργο εξαιτία των πάρα πολλών κυβερνοεπιθέσεων που είχε δεχθεί το τελευταίο διάστημα. Ξέρετε ότι ε, η υφιστάμενη κατάσταση μας καθιστά πιο ευάλωτους. Ξέρετε ότι προφανώς θα πρέπει να υπάρχουν τα δεδομένα διαθέσιμα για τις αρμόδιες αρχές, το επιχείρημα που χρησιμοποιείται πάρα πολύ για τις απαιτήσει εντοπισμού των εθνικών δεδομένων είναι ότι αν μια εταιρεία αποθηκεύσει δεδομένα σε ένα άλλο κράτος μέλος, μια αρμόδια εθνική αρχή δεν μπορεί να απαιτήσει τα δεδομένα αυτά και να έχει πρόσβαση σε αυτά. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να έχουμε και υψηλά πρότυπα κωδικοποίησης, κρυπτογράφησης για την προστασία των δεδομένων αυτών, έτσι ώστε να είναι ασφαλή εκεί που αποθεκεύονται. Προκειμένου όμως να στεφθεί με επιτυχία αυτή η πρόταση, είναι να μην επεκταθεί ο αριθμός των αποκλήσεων και των εξαιρέσεων. Θα πρέπει μόνο για λόγους δημόσιας ασφάλειας να επιτρέπονται εξαιρέσεις και παρεκκλήσεις. Αν αρχίσουμε να δίνουμε απλόχερα παρεκκλήσεις, τότε καταλαβαίνω ότι θα στραφούμε κατά της, ίδια, του ίδιου του στόχου της πρότασης αυτής. Σας ευχαριστώ πολύ και προσβλέπω στην καλή συνεργασία με τους υπόλοιπους συναδέλφους. Η κυρία Μούντι τώρα που αντικαθιστά τον κύριο Κόφωτ, όντως αντικαθιστώ τον κύριο Κόφωτ, ο συγητής για τους σοσιαλιστές, είναι σε μια άλλη σημαντική συνεδρία, δεν μπορεί να είναι εδώ και μου ζήτησε να μιλήσω εξ ονόματός του. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον συντάκτη μάλλον της για τις ε, σημαντικές σκέψεις τις οποίες μας ε, εξέθεσε και για το ότι ζήτησε να διοργανωθεί αυτή η πρώιμη ανταλλαγή απόψεων. Είμαι υπέρ τη πρωτοβουλία αυτή και θεωρώ ότι αναγκαία έρχεται την κατάλληλη στιγμή, καθότι όλο και περισσότερα κράτη-μέλη αρχίζουν και χρησιμοποιούν αδικαιολόγητα κριτήρια πρόσβαση στα δεδομένα του. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί πάρα πολλά εμπόδια και ένα μεγάλο άχθο για πολλέ επιχειρήσει και ιδίω για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Ξέρετε ότι για τις μεγάλες επιχειρήσεις το να υπάρχουν 20 ε, και πάνω τέτοια εμπόδια πρόσβασης στα δεδομένα είναι κάτι το επαχθές το οποίο καταφέρνουν όμως να ξεπεράσουν γιατί έχουν τα απαραίτητα μέσα. Δεν το καταφέρνουν όμως σε αυτό οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να δραστηριοποιηθούν διασυνοριακά γιατί δεν έχουν ε, τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους, ούτε την απαραίτητη τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, άρα δεν καταφέρνουν ε, να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και στους περιορισμούς τοπικοποίησης που θέτουν ορισμένα κράτη-μέλη. Άρα δεν μπορούν να δραστηριοποιηθούν πέρα από τα σύνορά τους. Ακριβώς λέει δηλαδή το αντίθετο από αυτό το οποίο θέλουμε να πετύχουμε στα, στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς. Αν θέλουμε μια γνήσια ενιαία εσωτερική αγορά θα πρέπει να καταρρύψουμε όλα αυτά τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν στην ελεύθερη ροή των δεδομένων. Μέσω της οδηγίας αυτής δεν θα πρέπει να περιπλέκουμε τα πράγματα περισσότερο από ό,τι ε, τώρα. Δεν έχει να κάνει πάντως με τα προσωπικά δεδομένα. Ξέρετε ότι υπάρχει η Γενική Οδηγία προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχουν επικαλύψεις ή αντιφάσεις ανάμεσα στις δύο αυτές οδηγίες. Θα ήθελα πάρα πολύ οι εκπρόσωποι τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μου δώσουν προς αυτό κάποιες διευκρινήσεις, έστω και γραπτός. Παράλληλα, νομίζω θα πρέπει να γνωρίζουμε πώς θα εφαρμοστούν στην πράξη όλοι αυτοί οι κανόνες για τα ιδιωτικά και μη ιδιωτικά δεδομένα. Θεωρητικά τα πράγματα μπορεί να είναι σαφή, στην πράξη όμως μπορεί να μην είναι τόσο εύκολο να υιοθετήσουμε τις δύο κατηγορίες. Ξέρετε ότι προφανώς οι επιχειρήσεις θα κληθούν να επεξεργάσουν και τις δύο κατηγορίες δεδομένων, άρα θα χρειαστεί να ανταποκριθούν σε δύο διαφορετικά νομοθετικά πλαίσια. Μπορεί και προς αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει κάποιες πληροφορίες. Και θα πρέπει βέβαια να πούμε προς τα κράτη-μέλη ότι θα υπάρχουν προφανώς και παρεκκλήσεις για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Παρ' όλα αυτά χρειαζόμαστε έναν καλύτερο ορισμό για το τι εννοούμε δημόσια ασφάλεια και οποιαδήποτε αφορά σε ζητήματα δημόσιας ασφάλειας δεν θα πρέπει να αποτελέσει μια απλή δικαιολογία προκειμένου να τεθούν περισσότεροι περιορισμοί τοπικοποίησης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρώιμη αυτή ανταλλαγή απόψεων και προσβλέπω στη συνεργασία με τους υπόλοιπους συναδέλφους. Ο κύριος Ντελούντε το λόγο ξανόματος των Πρασίνων. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα που θα συζητήσουμε και βεβαίως στη διάρκεια των συζητήσεων για την ολοκλήρωση και την υλοποίηση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, όπου θα έχουμε βεβαίως τη δυνατότητα να συζητήσουμε διάφορες διαστάσεις του ψηφιακού αυτού νέου κόσμου που δημιουργείται. Ένα ερώτημα όμως που πρέπει να απαντήσουμε από τώρα είναι ποιο, ποιο ακριβώς είναι το όριο, πώ οριοθετούνται τα προσωπικά από τα μη προσωπικά δεδομένα. Εδώ υπάρχουν διάφορες διατάξει, διάφορες δικαιοδοσίε και νομοθεσίες. Πώς θα εξασφαλίσουμε ότι θα ε, προστατεύεται η προσωπική ακαιρεότητα και η αξιοπρέπεια κάθε Ευρωπαίου πολίτη. Δεύτερον, διαλειτουργικότητα μεταξύ των ευρωπαϊκών συστημάτων. Εμείς ως πράσινοι θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να διευκολύνει την συνεργασία μεταξύ ε, υπαρχόντων αλλά και μελλοντικών παρόχων τεχνολογικών υπηρεσιών. Πάντως ε, χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση και βεβαίως σας διαβεβαιώνουμε ότι θα είμαστε ε, συμμέτοχοι ε, πάντοτε στη συζήτηση αυτή. Γιατί ο κύριος Ζαστανέ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Uh, in fact, Mr. Chair, my name is O'Donoghue, Director for uh, Future Networks. Uh, working uh, with uh, Pierre Είναι ο κύριος είναι ο διευθυντής. Ε, θα εκφραστούμε σύντομα από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από αυτή τη σύντομη συζήτηση προκύπτει ε, κάτι που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, ή μάλλον προκύπτει ότι τα μέλη γνωρίζουν πολύ καλά τους λόγους για αυτή την πρόταση και θα ήθελα να σταθώ σε λίγα σχόλια που ακούστηκαν και φυσικά περιμένουμε να συνεργαστούμε και με τα μέλη της Επιτροπής και με τον εισηγητή και το υπόλοιπο Κοινοβούλιο. Ισχύει ότι επίτηδες είναι μια βραχία πρόταση, μια σύντομη πρόταση τη Κομισιόν για να μην παρέμβουμε πολύ στην αγορά και για να κρατήσουμε την τεχνολογική ουδετερότητα. Προσπαθήσαμε λοιπόν να έχουμε κάποιε σαφείς νομικέ αρχέ, ορισμένε ακούστηκαν από εσά και τον εισηγητή και οι σκιώδεις εισηγητέ, για να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε ελεύθερη ροή δεδομένων. Δηλαδή, οι περιορισμοί που υπήρχαν ή που μπορεί να υπάρξουν στο μέλλον δεν θα επιτρέπονται για να δημιουργηθεί πραγματική ενιαία αγορά. Αλλά αυτό γίνεται όμως βάση, καταρχάς σαφών ρυθμίσεων σε ό,τι αφορά την κυβερνό ασφάλεια που δεν επηρεάζονται από αυτό, αλλά θα επηρεάσουν το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινούνται ελεύθερα και ρέουν ελεύθερα τα δεδομένα. Όπως είπαν και πολλοί ευρωβουλευτές, ένα βασικό θέμα ε, είναι ότι αυτό αφορά δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα. Μας ρώτησαν... Η... Μας ρώτησε η κυρία Μούντι από τους σοσιαλιστές να τις ε, πούμε συγκεκριμένα πράγματα γι' αυτό και σας διαβεβαιώνουμε ότι δεν υπάρχουν ε, επικαλύψεις, επικαλυπτόμενες διατάξεις και δεν υπάρχει περίπτωση παρεμβάσεων. Για να το εξασφαλίσουμε αυτό, έχουμε δώσει πρωτοκαθεδρία στον ε, Γενικό Κανονισμό προστασία ε, Προσωπικών Δεδομένων. Δηλαδή, οι ορισμοί που συμφωνήθηκαν από τους συνομοθέτες σε εκείνον τον κανονισμό που καθορίζουν το τι είναι προσωπικό δεδομένο, αυτό ισχύει υπεράνω όλων. Και μιλάμε για τα μη προσωπικά δεδομένα που υπόκειται σε αυτόν τον κανονισμό που συζητάμε τώρα. Ε, μπορεί να σα φαίνεται μια εύκολη λύση, αλλά δεν είναι. Προβλέψουμε τον κίνδυνο ότι αν είχαμε δύο διαφορετικούς ορισμούς, ένα για τα προσωπικά και τα μη προσωπικά δεδομένα, ε, υπήρχαν προβλήματα, εκτός και αν είναι απόλυτα ε, ευθυγραμμισμένοι. Στο μέλλον θα μπορούσαν να δημιουργηθούν τεχνικά προβλήματα. Ο ορισμός των μη προσωπικών δεδομένων στο γενικό κανονισμό μας επιτρέπει να λέμε ότι τα μη προσωπικά δεδομένα ε, είναι αυτά που δεν καλύπτονται από τον ορισμό εκείνου του γενικού κανονισμού. Γιατί το κάναμε αυτό, γιατί στο μέλλον θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ε, την τεχνολογία για να χρησιμοποιήσουμε ανώνυμα τμήματα δεδομένων ε, που αν τα συνδέσουμε, ας πούμε, μπορείς να εντοπίσει τον κάτοχο των δεδομένων. Προσοχή λοιπόν, προσοχή, προσοχή σε ό,τι αφορά τις τεχνολογικές εξελίξεις, σε ό,τι αφορά τον ορισμό της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Αυτός, αυτός απορρέει από την συνθήκη. Και υπάρχει και σχετική νομολογία που προήλθε από διάφορες υποθέσεις. Δεν θα σας κάνω μια πραγματεία τώρα, αλλά το δικαστήριο είπε ότι για να υπάρξει ε, δράση για την ε, δημόσια τάξη, αυτό προϋποθέτει την ε, ύπαρξη πραγματικής και σοβαρής απειλής που επηρεάζει τα βασικά συμφέροντα της κοινωνίας. Υπάρχει λοιπόν αυτή η νομολογία για να μας καθοδηγήσει ε, σε ποιο βαθμό δηλαδή, ο στόχος πολιτικής που αφορά την ασφάλεια θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ε, μέσω του περιορισμού των δεδομένων σε μια γεωγραφική περιοχή. Αυτά είναι κάποια από τα θέματα που θα τα δούμε μαζί, θα σας τα εξηγήσουμε, θα δώσουμε πληροφορίες και εξηγήσεις στην Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά τα παραδείγματα, φυσικά θα μπορούσαμε να δώσουμε κάποια παραδείγματα για τις δραστηριότητε παραδείγματο χάρη στον τομέα παραγωγή ενέργεια, αυτό που συζητούσατε προηγουμένω. Όπου παραδείγματο χάρη νημογεννήτριε που λειτουργούν τηλεματικό τρόπο και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα, φερρυπίν. Σε ό,τι αφορά, ας πούμε, όμως την ε, χρήση ε, ενέργειας από ένα άτομο, εκεί επειδή θα έχουμε, εκεί θα έχουμε προσωπικά δεδομένα, τιμολόγηση κτλ. Η Κομισιόν ξέρει ότι πολλές εταιρείες δεν θα είναι σε θέση αυτή τη στιγμή με ακρίβεια να λένε ποια από τα δεδομένα τους είναι προσωπικά και ποια δεν είναι προσωπικά. Συχνά αποθηκεύονται και τα μέ και τα δε ε, είτε στο ίδιο hardware ή στον ίδιο υπολογιστή, στον ίδιο χώρο. Αλλά η στο ιδιο υπολογιστη στον ιδιο χωρο αλλα η προστασια των προσωπικών δεδομένων ισχύει. Αν υπάρχουν αμφιβολίες, αν υπάρχουν ας πούμε ίχνη προσωπικών δεδομένων σε μια δέσμη δεδομένων, θα πρέπει να προστατεύονται με βάση τους κανόνες προστασίας ε, προσωπικών δεδομένων. Αυτά είναι θέματα που υπάρχουν ε, και εξετάζονται από το Συμβούλιο. Με μεγάλη χαρά βέβαια θα σας δώσουμε περαιτέρω εξηγήσεις και πληροφορίες, καθώς θα εξελίσσονται εδώ οι συζητήσεις στο Κοινοβούλιο. Και να κλείσω, Πρόεδρε, λέγοντας ότι είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο, ούτως ώστε μαζί τα θεσμικά όργανα να μπορέσουν να υλοποιήσουν τους στόχους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ε, στην ε, ε, Σύνοδο για τα ψηφιακά θέματα πριν από τρει-τέσσερι εβδομάδε, όπου ζήτησαν του συνομοθέτε να προσπαθήσουν να υιοθετήσουν αυτόν τον κανονισμό μέχρι τα μέσα του 18 το αργότερο. Ε, περιμένω και προσβλέπω στη συνεργασία μα. Πολύ ωραία. Ο Κάσνοντεύσκη, ο εισηγητή μα ακόμα μια φορά. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Και νομίζω ότι όλα αυτά τα θέματα θα χρειαστεί να τα συζητήσουμε στη διάρκεια των συνεδριάσεων των ε, σκιωδών προκειμένου να δούμε κατά πόσο μπορούμε να βελτιώσουμε περαιτέρω αυτήν την εξαιρετική γνωμοδότηση. Και ελπίζω να προχωρήσουμε γρήγορα με τη διαδικασία των τροπολογιών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ωραία. Μεγάλη πειθαρχία έχουμε επιδείξει και έχουμε κάποιο χρονικό περιθώριο κερδίσει χάρη σε αυτή την πειθαρχία και μπορούμε να περάσουμε στην, ε, στην ε, συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βραζιλίας σε θέματα επιστημονικού ενδιαφέροντος. Να σας υπενθυμίσω ότι το, η συμφωνία αυτή αφορά την τεχνολογική και επιστημονική συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Βραζιλίας. Έχουμε ε, δεσμεύσει, σχεδιάσει να κάνουμε μια δεκάλεπτη συζήτηση. Θα ήθελα ο κύριος Τσιόκα να μας παρουσιάσει την θέση του. Έχετε τρία λεπτά στη διάθεση σας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, τις επόμενες μέρες θα λάβετε το κείμενο που αφορά την ανανέωση της Συμφωνίας Συνεργασίας Επιστημονικής και Τεχνολογικής Φύσεως μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας. Η συμφωνία Ισχύει από το 2007 μέχρι σήμερα και από το 2007 μέχρι σήμερα επέτρεψε να σημειώσουμε πρόοδο σημαντική σε ό,τι αφορά την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία. Η συνεργασία μεταξύ των ερευνητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Βραζιλιάνων ερευνητών μας επέτρεψε να φέρουμε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Είναι σημαντικό σήμερα να συνεχίσουμε σε αυτό τον δρόμο, να μην χαλαρώσουμε και να μην διακόψουμε αυτή την ε, συμφωνία. Γι' αυτούς τους λόγους θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υποβάλω στους συναδέλφους ε, την ανανέωση για πέντε χρόνια αυτής της συμφωνίας που θα μας επιτρέψει να εξακολουθούμε να έχουμε σημαντικά αποτελέσματα και να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βραζιλίας, κυρίως στους τομείς προτεραιότητας της επιστήμης και της τεχνολογίας. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για την προσοχή τους και σας ευχαριστώ και σας κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Μπουζόητορ για το έλικα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον εισηγητή. Νομίζω ότι είναι πολύ θετική συμφωνία αυτή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο τομέας της έρευνας ε, τομείς κοινού συμφέροντος όπως η βιοινφορματική, η νανοτεχνολογία, η έρευνα, οι καθαρές πηγές ενέργειας, η βιοασφάλεια, η υγεία και η ιατρική είναι πολύ σημαντικοί τομείς και πολύ σημαντικά ζητήματα όπου θα μπορούσαμε πραγματικά να υποφεληθούμε από τις αμοιβέ αυτές ερευνητικέ δραστηριότητες και από την αμοιβαία πρόσβαση στην τεχνολογία που προβλέπει αυτή η συμφωνία. Το ΕΛΚ λοιπόν υποστηρίζει την ανανέωση της συμφωνίας αυτής για πέντε ακόμα χρόνια, όπως συμφώνησαν στην αρχή του έτους και τα συμβαλόμενα μέρη. Ο στόχος είναι να ενθαρρύνουμε και να διευκολύνουμε τη συνεργασία των συμβαλωμένων μερών και στους τομείς αυτούς, αλλά και σε άλλους τομείς κοινού συμφέροντος και να καταφέρουμε τελικά να έχουμε περισσότερες τεχνολογικές και επιστημονικές κοινέ δραστηριότητες και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επωφελείται σφαιρικώς. Δεν βλέπω λοιπόν για ποιο λόγο να μην υποστηρίξουμε την ανανέωση της εν συμφωνίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ζωρίνιο τώρα έχει το λόγο για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σιγητά, αγαπητοί συνάδελφοι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρότεινε την αναθεώρηση, την ανανέωση μάλλον, της Συμφωνίας Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βραζιλίας για πέντε ακόμα χρόνια. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ λογική η πρόταση αυτή, το πάνε και οι συνάδελφοι, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να υποστηρίξει αυτή την ανανέωση. Η συμφωνία αυτή αποτελεί πολύ σημαντικό σημείο αναφοράς για την ε, μεταφορά τεχνογνωσίας και γνώσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βραζιλίας. Εγώ είμαι αντιπρόεδρος της ε, αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τη Βραζιλία. Είχα πάει πρόσφατα στη χώρα αυτή και μπορώ να σας πω πραγματικά ότι υπάρχουν απτά αποτελέσματα από την τεχνολογική και επιστημονική αυτή συνεργασία. Είμαστε δύο εταίροι οι οποίοι πραγματικά συνεργαζόμαστε πάρα πολύ αποτελεσματικά. Υπάρχει ένας φορέας στη δική μου τη χώρα, την Πορτογαλία, όπου συνεργάζεται στον τομέα της αεροναυπηγικής με αντίστοιχο φορέα από τη Βραζιλία τέτοια συνεργασία και τέτοιες συνεργασίες θεωρώ ότι γίνονται ακόμα πιο σημαντικές αν καταφέρουν τελικά σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα να επωφελούνται και από μια συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μερκοσούρα. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης, καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τους πολίτες και θεωρώ ότι η συμμετοχή της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το Σύντρα, για παράδειγμα, στην Πορτογαλία και τον αντίστοιχο φορέα που υπάρχει στη Βραζιλία, από την άλλη πλευρά δηλαδή του Ατλαντικού, δίνει μια περαιτέρω όθηση στη συμφωνία αυτή. Η ε, δήλωση που έγινε στην ε, Λισαβόνα καταδεικνύει τελικά ότι μιλάμε εδώ πέρα για μια συμφωνία επιστημονική και τεχνολογική που ασχολείται με ζητήματα όπως οι κλιματικές αλλαγές, τα ρεύματα στους ωκεανούς και το καθεξής. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ανανεώσουμε τη συμφωνία αυτή και ως σοσιαλιστές υποστηρίζουμε την πρόταση του Συμβουλίου. Σας ευχαριστούμε κύριε Ζωρίνιο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που λειτουργείτε ως γέφυρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βραζιλίας. Ο κύριος Τσέζεκ τώρα έχει το λόγο εξ του ΙΣΙΑΡΑ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή για τη σύντομη παρουσίαση που έκανε και να ευχαριστήσω και όλους τους αδέρφους που πήραν το λόγο πριν από μένα. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να πω ότι είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο με την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βραζιλίας σε αυτόν τον τομέα. Βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της υποστηρίζουν ε, τη δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να δούμε λίγο πέρα από τα δικά μας τα σύνορα και να καταφέρουμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας και με άλλες χώρες. Όπως είπε και ο συνάδελφος από το ΕΛΚΑ, θα ήθελα και εγώ να πω ότι η Βραζιλία είναι ανάμεσα στις πιο σημαντικές χώρες όσον αφορά την έρευνα που γίνεται στο γεωργικό τομέα και συγκεκριμένα στα βιοκαύσιμα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει και στον τομέα αυτό να επεκτείνουμε λίγο τη συνεργασία μας. Νομίζω ότι είναι απόλυτα δικαιολογημένο να ενσωματωθεί και αυτός ο τομέας στο τελικό σχέδιο εντολής για τη συμφωνία αυτή. Και ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα καταφέρει σύντομα να διεκπαιρώσει το φάκελο αυτό προκειμένου όντως να νεωθεί η συμφωνία αυτή και να καταφέρουμε και εμείς να υποστηρίξουμε την ήδη πολύ θετική συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βραζιλίας, η οποία όπως είπα είναι αμοιβαία αποφελής. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε πολύ. Να ζητήσω τώρα από τον κύριο Τσόκα να απαντήσει σε αυτές τις παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους οι οποίοι τόνισαν πόσο σημαντική είναι η συμφωνία αυτή, πόσο σημαντικό να καταφέρουμε να συνεχίσουμε την εργασία αυτή που έχει ξεκινήσει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βραζιλίας. Αναφέρθηκαν κάποια σημεία τα οποία θεωρώ ότι είναι σημαντικά και τα οποία θα πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη στα πλαίσια του κειμένου που επεξεργαζόμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στις εργασίες μας. Ευχαριστούμε πολύ. Να σας ε, ενημερώσω ότι η ημερομηνία κατάθεσης τροπολογιών είναι 14 Δεκεμβρίου. Θα περάσουμε τώρα στο τελευταίο σημείο της ε, ημερήσιας διάταξης που ήταν τόσο φορτωμένη για σήμερα το απόγευμα. Μελέτη σχετικά με την επανεξέταση της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών ε, ε όσον αφορά πολιτικές που επιπτούν στον τομέα δραστηριοτήτων της Ήτρας σε σχέση με το Brexit. Παρουσίαση από τον κύριο Σκοτ Μάρκους ε, που είναι μέλος του Think Tank Brugge που έχει, παρουσιάσει, που έχει προετοιμάσει και μια παρουσίαση για εμάς. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Λοιπόν, μια και έχουμε κερδίσει λίγο χρόνο σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα, καλό θα είναι να το διατηρήσουμε αυτόν τον χρόνο για να έχουμε ε, περισσότερο χρόνο για να προχωρήσουμε σε συζήτηση και ερωτήσει μετά. Λοιπόν, Ας αξιοποιήσουμε τον χρόνο που έχουμε τώρα ε, για να περάσουμε στο τελευταίο θέμα. Η επόμενη ε, συνεδρίασή μας θα γίνει 7 ε, Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί. Θα είναι κοινή συνεδρίαση με την ΕΝΒΗ και θα ψηφίσουμε και επί του θέματος της διακυβέρνησης. Και μετά έχουμε συνεδρίαση 11 Ιανουαρίου από τις 9 έως τις 12.30 εδώ στις ε, Βρυξέλλες και η, η αρχική συνεδρία ήταν προγραμματισμένη να γίνει 11 Δεκεμβρίου. Ε, αυτή έχει ακυρωθεί. Αυτό συμφωνήθηκε σήμερα το πρωί στην ε, συνάντηση των συντονιστών. Ελπίζω λοιπόν ε, ότι στο μεταξύ έχει καταφτάσει και ο προσκεκλημένος ομιλητής μας. Δεν ξέρω να κοιτάξω. Where is the study we, uh, he will talk about? Uh, all of us will... Αυτή είναι η μελέτη. Θα λάβετε όλοι αντιγράφω αν δεν έχετε λάβει ήδη. Με κάποια εισαγωγικά λόγια, ούτως ώστε να έχουμε και πιο σύντομη παρουσίαση. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε αυτή την έκθεση που ετοιμάστηκε το πρώτο μισό του 2017 και όπου προσπαθούμε να δούμε τους διάφορους ε, τομείς ε, που ε, απασχολούν την Ήτρε, ανάπτυξη, της, ανάπτυξη έρευνα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενέργεια, περιβάλλον, ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Προσπαθήσαμε να αναλύσουμε ποια μοντέλα υπάρχουν για συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών ούτως ώστε για κάθε μοντέλο να εντοπίσουμε για δύο χώρες, Νορβηγία με την ε, ε, Ελβετία, με ιδιαίτερες ε, διμερείς σχέσεις, Ουκρανία, μέλος της ενεργειακής κοινότητας, που έχουν πολύ ενδιαφέρουσα δέσμη κανόνων που τη συνδέουν αυτές τις χώρες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. για το ερευνητικό κομμάτι μπορείς να πεις εσύ δύο-τρία πράγματα. Εσείς ξέρετε ποιος είναι ο καλύτερος, ο πιο αρμόδιος για να μας μιλήσει για το κάθε θέμα. Here he is. Κύριε Μάρκους, σας περιμέναμε. Τελειώσαμε νωρίτερα. νωρίτερα. Δεν είναι δικό σας λάθος. Δεν έχετε καθυστερημένος. Ζητώ συγγνώμη. Νόμιζα ότι είχα χρόνο. Παρακαλώ ανεβάστε τις φωτοτυπίες, τις α, συγγνώμη. Ωραία. Καταρχάς, χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ. Είναι μια μελέτη που εκπονήσαμε για την Επιτροπή ΙΤΡΕ, για το Τμήμα Πολιτικής. Την ολοκληρώσαμε την Άνοιξη, τη δημοσίασαμε την Άνοιξη και μαζί μου σήμερα ε, έχω δύο από τους συναδέλφους από τον Μπρούγκελ, τον κύριο Φρέγκλερ Φρέγκλερς που είναι ε, ερευνητής, ειδικός ερευνητής και τον κύριο Ζάκμαν που είναι ε, εμπειρογνώμονα σε θέματα περιβάλλοντος και ενέργειας και ο οποίος συμμετείχε και σε μια άλλη μελέτη η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα και αφορά τις επιπτώσεις του Brexit στο σύστημα ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ίδια η μελέτη λοιπόν ε, αξιολογεί υπάρχοντα μοντέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες, δηλαδή χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μελέτη λοιπόν εκπονήθηκε από την σκοπιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιλέξαμε να μην ε, ε, ε, εικάσουμε τι θα ήθελε ή τι θα επιδίωκε το, το Βασίλειο. Κοιτάζουμε τα θέματα αυτά από σκοπιά Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η, ιδιότητα του μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης λοιπόν αποτελεί τη βάση μας, η ιδιότητα του μέλους του ΕΟΧ, ε, Υπάρχουν ε, από εκεί και πέρα βεβαίως διμερείς ε, διευθετήσεις και συμφωνίες με κράτη της ΕΖΕΣ, μιλώ για την ελβετική περίπτωση και υπάρχουν και άλλα μοντέλα. Είναι τέσσερις οι θεματικές κατηγορίες που εξετάσαμε. Ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ενέργεια και περιβάλλον, ερευνητική πολιτική και ε, μικρές επιχειρήσεις. Αυτές είναι οι αρμοδιότητές σας. Δεν κάνουμε συστάσεις, προσπαθούμε να συλλέξουμε κάποιες ε, πληροφορίες προκειμένου να μπορείτε να λαμβάνετε τεκμηριωμένες αποφάσεις. Ας μιλήσουμε λοιπόν για τα τρία διαφορετικά μοντέλα. Ε, μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέλος του ΕΟΧ και ε, διμερείς διευθετήσεις και συμφωνίες, ελβετικό μοντέλο δηλαδή. Στην περίπτωση των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι χρειάζεται να κάνει είναι προφανώς ε, η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Κάθε κράτο μέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζει το σύνολο της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Ε, παρόμοια είναι τα πράγματα στην περίπτωση των μελών του ΕΟΧ, κάποια όμως θέματα ε, εξαιρούνται, ε, όπως για παράδειγμα η Αλία και η Γεωργία. Στην ελβετική περίπτωση υπάρχουν δεκάδες διμερείς συμφωνίες και υπάρχουν και κάποιοι κανόνες, κάποιοι τομείς που δεν ρυθμίζονται καθόλου, άλλοι τομεί που ρυθμίζονται με μεγάλη λεπτομέρεια. Αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι πώς θα καταφέρουμε ε, να επιτύχουμε τις απαιτούμενες αλλαγές στο ευρωπαϊκό κεκτημένο με την πάροδο του χρόνου. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν οι οδηγίες θα πρέπει, πρέπει να μεταφέρονται στο Εθνικό Δίκτυο των Κρατών Μελών. Ε, το ίδιο ισχύει και για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ενώ στην περίπτωση της Ελβετίας μπορούν να ε, συναυθούν νέες συμφωνίες χωρίς να υπάρχει όμως συγκεκριμένος ε, μηχανισμός όσον αφορά την ε, προσαρμογή του ελβετικού δικαίου με βάση τις αλλαγές που γίνονται στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Εδώ λοιπόν εξετάζουμε το ζήτημα της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Αν δείτε τη μελέτη και το ενημερωτικό σημείωμα περιλαμβάνει πάρα πολλούς πίνακες και διαγράμματα προκειμένου να καταστούν οι πληροφορίες που συλλέξαμε πιο κατανοητές στους αναγνώστες. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι το, Ευρωπαϊ... το Βασίλειο είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και έχει υπάρξει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρόσφατο παρελθόν. Θέλαμε λοιπόν να ε, χρησιμοποιήσουμε το Ηνωμένο Βασίλειο ως ε, παράδειγμα προκειμένου να ξάγουμε τα σημαντικότερα, τα, καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, ε, συμπεράσματα με βάση ε, την περίπτωσή του. Το Ηνωμένο Βασίλειο λοιπόν εφαρμόζει πλήρως την νομοθεσία. Η Νορβηγία μαζί με την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν είναι τα μέλη του ΕΟΧ. Και εδώ υπάρχει μια ε, σε μεγάλο βαθμό εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου, όχι πλήρης όσον αφορά την έννοια αγορά, αλλά ε, δεν, δεν, υπάρχει ε, ε, ακόμη και όταν δεν κατοχυρώνεται νομοθετικά η προσαρμογή του νορβηγικού δικαίου στο ευρωπαϊκό υπάρχει μεγάλο επίπεδο συντονισμού. Στην περίπτωση της Ολυβητίας όσον αφορά την εφαρμογή των πολιτικών της ενιαίας αγοράς εκεί τα πράγματα είναι κάπως αδύναμα. γιατί, για παράδειγμα, δεν εφαρμόζονται οι κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης στο φυσικό αέριο στην Ελβετία δεν υπάρχει συγκεκριμένος μηχανισμός θέσης στόχων, υπάρχει ένας συντονισμός χωρίς ωστόσο να υπάρχει ε, νομική δεσμευτικότητα. Στην ε, Ουκρανία υπάρχει και εδώ μια εν μέρη εφαρμογή, ιδίως όσον αφορά τους κανόνες ε, για, για το κλίμα, το περιβάλλον και τον ενεργειακό εφοδιασμό και την ασφάλειά του. Αυτός ήταν ένας από τους τέσσερις τομείς. Αν δούμε τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, εδώ βλέπουμε ότι η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνέβαλε πολύ προκειμένου να ε, ενισχυθεί η εναρμονισμένη εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Πρόκειται για ε, έναν από τους τομείς κλίμακας για το Ηνωμένο Βασίλειο και αποτέλεσε και έναν παράγοντα σύγκλησης ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δείτε την Νορβηγία ως παράδειγμα του μέλους του ΕΟΧ, βλέπουμε ότι υπάρχουν περίπου τα ίδια πλεονεκτήματα από τη συμμετοχή της χώρας στον ΕΟΧ. Οι διμερείς συμφωνίες στην Ελβετία σε σχέση με τη συμμετοχή μιας χώρας στον ΕΟΧ ε, έχουν αποδειχθεί λιγότερο αποτελεσματικές όσον αφορά την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου και, και όσον αφορά την σύγκληση. Οι χρεώσεις περιαγωγής είναι υψηλότερες στην Ελβετία, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, αλλά και οι ρυθμοί ε, ε, ε τερματισμού καταγγελίας ε, τηλεπικοινωνιακών συμβάσεων στην, στην, Ευρωπαϊκή, στην ε, Ελβετία είναι πάρα πολύ υψηλές ιδίω σε σχέση με τα, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα το σύστημα δεν απέφερε ιδιαίτερα αποτελέσματα όσον αφορά την οικονομική σύγκληση της Ελβετίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ε, εξετάσαμε το ζήτημα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στις ε, Συμφωνίες Ελευθέρων Συναλλαγών και έχουμε εδώ τέσσερις περιπτώσεις συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν είναι ότι στην ε, συμφωνία με την Νότια Κορέα, σε αυτές τις νέες συμφωνίες έχουν επιτευχθεί υψηλά επίπεδα πρόσβαση στην αγορά. Ωστόσο, ε, το σχέδιο δεν, ήταν ποτέ, δεν περιλάμβανε ποτέ ρυθμιστική σύγκληση. Κινούνται γύρω από την αρχή της μη διάκρισης και της πρόσβασης στην αγορά οι συμφωνίες ε, ελευθέρωσης στην αγορά. Οπότε δεν απέφεραν πολλά αποτελέσματα όσον αφορά τη σύγκληση, τη ρυθμιστική. Όσον αφορά την ερευνητική πολιτική, βλέπουμε ότι το πρόγραμμα ορίζοντα 2020 είναι το βασικό εργαλείο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως και τα προηγούμενα πλαίσια, ε, προγράμματα πλαίσιο, είναι το βασικό εργαλείο. Ε, Υπάρχουν βεβαίω και μορφέ συνεργασία με χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συνδεδεμένε χώρε, ή οντότητε ε, τρίτων χωρών ε, απολαμβάνουν ε, το ίδιο καθεστώς σε μεγάλο βαθμό με, τα, με τις οντότητες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επιλέξιμες ε, οντότητες από τρίτες χώρες, αλλά ακόμη και, και χώρες οι οποίες έχουν ε, διμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το Ισραήλ. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νορβηγία και η Ελβετία δέχονται χρηματοδότηση εποφελούνται από τη, από τη και βεβαίω από τη συνεργασία με τα ερευνητικά κέντρα που προωθεί και υποστηρίζει το πρόγραμμα ορίζοντα 2020. Αν δούμε τώρα τι μικρέ επιχειρήσει, το βασικό εργαλείο είναι το πρόγραμμα COSME, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή από το 2014. Δεν περιλαμβάνει πάρα πολύ μεγάλα ποσά, αλλά τα ποσά αυτά ε, χαρακτηρίζονται από υψηλή μόχλευση. 65% ε, των χρημάτων πηγαίνουν σε εγγύησει δανείων για μικρέ και μεσέ επιχειρήσει και ε, με αυτόν τον τρόπο ε, αυξάνεται η ιδιωτική ε, χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Εδώ η πρόσβαση αφορά κράτη-μέλη, κράτη-μέλη του ΕΟΧ. Δεν συμμετέχουν όμως όλα τα κράτη-μέλη. Η Ισλανδία συμμετέχει ε, η Νορβηγία και το Λιχτενστάιν δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα κόσμου. Πάντως η ιδιότητα του μέλους είναι ανοιχτή σε όλα τα κράτη όπου φάνηκε ότι υπάρχει ενδιαφέρον ε, προκειμένου να προωθηθούν οι μικρές επιχειρήσεις. Υπάρχουν και άλλα εργαλεία που αφορούν την επιχειρηματικότητα, την, ε, κατάρτιση καθώς και τη, τη διάθεση στη διεθνή αγορά των προϊόντων και εμπορευμάτων. Πάντως το κόσμο προωθεί αυτή την ε, συνεργασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι τα βασικά πορίσματα λοιπόν. Το πρώτο είναι ότι ε, θεωρώντας ότι το ε, Ηνωμένο Βασίλειο πράγματι θα αποχωρήσει υπάρχουν τέσσερις τομείς ε, όπου αποδεικνύεται ότι από σκοπιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, η ιδιότητα του μέλους του, ή το μοντέλο του, του μέλους του ΕΟΧ θα είναι εκείνο που θα εξασφαλίσει τα μεγαλύτερα ωφέλη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, η συμμετοχή στον ΕΟΧ ε, ενισχύει ε, τον, τη σύγκληση. Είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή όσον αφορά την συνέπεια των νομοθετικών πλαισίων, το βαθμό της οικονομικής σύγκλησης αλλά και της ρυθμιστικής σύγκλησης. Η συμμετοχή στην ενεργειακή κοινότητα, όπως, κάνει, όπως, ε, αφορά, όπως ισχύει στην περίπτωση της Ουκρανίας, μπορεί να βοηθήσει στην εναρμόνιση των ε, νομοθεσιών. Αλλά υπάρχουν και κάποιες, κάποιοι περιορισμοί. Οι κανονισμοί ε, εναρμόνισης μπορεί να είναι δύσκολο να εφαρμοστούν στην πράξη, συμβάλλει θετικά στη σταθερότητα και την ασφάλεια του εφοδιασμού, συμβάλλει θετικά στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, αλλά φαίνεται ότι είναι λίγο αποτελεσματική όσον αφορά την εξασφάλιση δίκαιης πρόσβασης στην αγορά για τις ευρωνοσιακές επιχειρήσεις. Αυτό είναι ένα από τα βασικά μας πορίσματα. Όσον αφορά την, το μοντέλο ε, FTA, λαμβάνοντας υπόψη ως παράδειγμα το, την Νότια Κορέα και αυτή αποφέρει θετικά αποτελέσματα, ωστόσο αποφέρει μικρά θετικά αποτελέσματα ε, σε ρυθμιστικά ζητήματα. Αλλά και αυτά όχι ε, αμεληταία, ε, καθώς για παράδειγμα δεν υπήρχαν στην Κορέα ούτε στη συμφωνία ε, που υπογράφηκε με την Κορέα συγκεκριμένε διατάξει για την αγορά χονδρική. Παρ' όλα αυτά, η Κορέα από μόνη τη αποφάσισε να θεσπίσει σχετικού κανόνε. Όσον αφορά το κόσμο και το ορίζοντας 2020, ε, το βασικό ερώτημα είναι ε, πώς θα εξασφαλιστεί συμμετοχή αλλά και αμοιβαίο όφελος. Αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει είναι μας ενδιαφέρει πλέον να, ε, να χρηματοδοτούμε οντότητες επιστημονικούς ερευνητικούς φορείς σε χώρα η οποία δεν θα συμμετέχει πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός, αυτή είναι η μεγάλη μεταβλητή, το μεγάλο ερωτηματικό. Αυτά ε, ε, έχουμε και πάρα πολύ χρόνο πλέον αφού εγώ ολοκλήρωσα για να ακούσουμε ερωτήσεις και να προχωρήσουμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση αν θέλετε. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Υπάρχουν ερωτήσεις κυρία Μούντι surprise, the British MEP in the room <laughs> some Είμαι ο μόνος ε, Βρετανός ε, πολιτικός στην αίθουσα. Τι περίεργο. Σας ευχαριστώ για τη μελέτη. Και εγώ πιστεύω ότι το καλύτερο μέλλον ε, για το Ηνωμένο θα ήταν να μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, για να ξεκαθαρίσουν τις παρεξηγήσεις. Αλλά αν δεν συμβεί, έχω κάποιες ερωτήσεις για πράγματα που δεν είπατε που είναι και τομείς που απασχολούν την Επιτροπή μου. Τουλάχιστον δεν τα αναφέρατε στις διαφάνειές σας. Όταν, αναφέρουμε, όταν κοιτάμε το τομέα της έρευνας, αυτό που δεν είπατε είναι τι γίνεται με το Εράσμους. Και το τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας, που είναι τεράστια ανησυχία, τεράστιο μέλημα και η συνεργασία ξεπερνάει τα προφανή. Κάτι που δεν αναφέρατε, δεν ξέρω αν μιλήσατε για το διάστημα καθόλου, που είναι εντολή, το, δηλαδή είναι αρμοδιότητα της δική μας Επιτροπής. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι για το θέμα του διαστήματος. Για το κεφάλαιο της ενέργειας, επίσης, επίσης ε, δικό μας, δική μας αρμοδιότητα, είναι, αφορά τη σύνδεξη, τη συνεργασία για τη σύνδεξη, είπε για τη Euratom. Τι πετύχαμε ε, πραγματικά και τι θεωρητικά, ας πούμε. Είναι σημαντική διάφορα για να μην ξεχάσουμε κάτι και κυρίως ε, ορισμένοι παραπλανηθούν. Άλλε ερωτήσει. υπάρχουν. Ακούσαμε από την κυρία Μούντι ότι κατά την άποψή τη το Brexit είναι επιζήμιο για το Ηνωμένο Βασίλειο. Για μένα είναι τουλάχιστον το ίδιο επιζήμιο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω πρόβλημα τώρα με οργανισμούς όπως ο δικός σας που εκφράζουν ουδέτερη άποψη. Δεν παίρνουν θέση. Έχει περάσει μισό χρόνος από το δημοψήφισμα και τώρα οι Βρετανοί αρχίζουν να συνειδητοποιούν τι σημαίνει το Brexit. Αλλά δεν νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι έχουν συνειδητοποιήσει τι σημαίνει για την Ευρωπαϊκή Ένωση το Brexit. Αν κοιτάξετε τον ορίζοντα 2020, να ένα θαυμάσιο αποτέλεσμα της καταστροφικής συνέπειας του Brexit. Αν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι πια εταίρος, θα είχαμε πρόβλημα. Ακούσαμε από πολλούς εδώ στις Βρυξέλλες ότι μια χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι η προαναγγελία μιας τιμωρίας. Γιατί μην ξεχνάμε το Ισραήλ, ας πούμε, που έχει την ίδια μεταχείριση με χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, η πρώτη μου ερώτηση είναι γιατί Εν τη αυτή περιπτώσει, το Ηνωμένο Βασίλειο να μην έχει την ίδια μεταχείριση με το Ισραήλ, που δεν είναι καν ευρωπαϊκή χώρα. Ούτε καν τη Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώ. Και δεύτερον, ε, ένα φορέα όπω ο δικό σα, που εξετάζει τι έχει συμβεί στο παρελθόν ε, γιατί μας παρουσιάσετε τώρα τη μελέτη σας. Ε, δεν θα, είχε νόημα να παρουσιάσετε τη μελέτη σα πριν το δημοψήφισμα ούτως ώστε να ξέρουν οι Βρετανοί τι νόημα έχει για αυτού και τι συνέπειε έχει για αυτού το Brexit. Και κάτι άλλο που δεν αφορά την ήτρα και τι αρμοδιότητέ τη, αλλά έρχεται στο μυαλό μου. Το θέμα τη μετανάστευση. Έχει αλλάξει η στάση τη ε, Ευρώπη. Τώρα για, για σας, για την οργάνωσή σας, δεν θα, ήταν, δεν θα είχε νόημα να πείτε αυτή η συζήτηση για ήπιο ή σκληρό Brexit δεν έχει κανένα νόημα. Εσείς ε, λέτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα. Ποιος πρέπει να προτείνει αυτή την αλλαγή. Εσείς αν μα ρωτάτε ποιο είναι ο ρόλος τη της μα μας οργάνωσης, αυτό που σας παρουσίασα είναι μια μελέτη που έγινε για το δικό σας policy department. Σε αυτή τη μελέτη ε, εμείς ε, παρουσιάζουμε τα πράγματα με ουδετερότητα. Αν κοιτάξετε άλλες θέσεις που έχουμε πάρει εμείς τα, τελευταία δύο χρόνια, τότε οι συνάδελφοί μου με συνέπεια είπαν, πιστεύουμε, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα... ήταν καλό να παραμείνει. Επίσης λέμε ότι η σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι σημαντική και δεν θα πρέπει να υποβαθμιστεί περισσότερο από ό,τι χρειάζεται σαν αποτέλεσμα του Brexit. Ε, φεύγουμε του πεδίου της μελέτης, αλλά η δική μου οργάνωση ήταν πάντα πολύ συνεπή στο τι λέει. Και η δική μου άποψη ίδια είναι. Πιστεύω ότι το δημοψήφισμα ήταν ατυχές. Πιστεύω ότι οι συνέπειες θα είναι πολύ μεγαλύτερε Έτσι, προσωπική άποψη. Δεν είναι και τόσο ριζοσπαστική. Η επίπτωση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη για τον Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρώπη. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πολύ μεγαλύτερο ε, εμπορικό, ας πούμε, έχει πολύ μεγαλύτερο εμπορικό βάρος από το Ηνωμένο Βασίλειο. Παρ' όλα αυτά είναι επιζήμιο και για τους δύο. Ίσως ε, δεν καταλάβαμε την πρόθεση, αλλά όταν ε, δουλεύουμε με λογαριασμό του Policy Department, ε, στην πραγματικότητα εκφράζουμε την άποψή μας με ουδετερότητα. Καταλαβαίνω τι μου λέτε εσείς τώρα και συμφωνώ ότι η έκθεση όπως έχει είναι ουδέτερη. Προσπαθεί να είναι ουδέτερη ούτως ή άλλως. Ίσως θα μπορούσε να έχει, πάει, να έχει κινηθεί σε άλλη κατεύθυνση. Σε ό,τι αφορά τις αρχικές ερωτήσεις που ακούσαμε από την κυρία Μούντι αφορούν διάφορους τομείς για το διάστημα. Δεν μας το ζήτησαν να το κοιτάξουμε και δεν το κοιτάξαμε. Δεν υπάρχει ούτε σε αυτήν την έκθεση ούτε στην επόμενη ε, που ασχολείται με τις επιπτώσεις στο ενεργειακό σύστημα. Σε ό,τι αφορά το έρασμους και το θέμα της ε, ελεύθερης κυκλοφορίας των ακαδημαϊκών. Θα μιλήσει η συνάδελφος και για το θέμα της ενέργειας και της σύνδεξης ο Γκέοργ μπορεί να πει κάτι. Γιατί αφορά και την έρευνα και την ενέργεια το ζήτημα αυτό. Η συνάδελφος πρώτη θα μπορούσε να μιλήσει για το Εράσμους και το θέμα της ελεύθερης κυκλοφορίας. Στον τομέα της έρευνας. Μιλάμε για την ελεύθερη κυκλοφορία των ερευνητών, που ήταν βασικό στοιχείο του, χώρου, του ερευνητικού χώρου της ενέργειας η κυκλοφορία δεν είναι μόνο το Εράσμους, που είναι σημαντικό τμήμα βέβαια, αλλά έχουμε και το μαρίκιουρι Κιουρί για τους μεταδιδακτορικούς φοιτητέ. Το Εράσμος είναι σημαντικό κομμάτι φυσικά. Αυτό που λέει η έκθεσή μας είναι ότι αυτή η κυκλοφορία είναι πάρα πολύ σημαντική και τις δύο πλευρές. Ε, βελτιώνει την, ε, το επίπεδο της επιστήμης συνολικά. Και ο ορίζοντας 2020 επιτρέπει λοιπόν την ελεύθερη κυκλοφορία. Ε, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι όχι μόνο το, η περίπτωση της Ελβετίας, αλλά όπου συνειδητοποιήθηκε ότι μειώντας την ε, κινητικότητα, μειώνεται η αποτελεσματικότητα χάνουν οι Ελβετοί, αλλά χάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ελεύθερη κυκλοφορία, η κινητικότητα είναι βασικό στοιχείο, προϋπόθεση ούτω ώστε να επωφεληθούμε από την, ερευνητική, από την Ευρωπαϊκή Ερευνητική Περιοχή. Για το διάστημα τώρα. Σε κάποιο βαθμό, ναι, είναι τμήμα του ορίζοντα 2020, αλλά τα νέα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εκφεύγουν του ορίζοντα 2020 και θέτουν το διάστημα σε διαφορετική βάση. Η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντική. Γιατί ανάλογα με το που ανήκεις μπορεί να συμμετάσχεις πλήρως στη συζήτηση Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διάστημα αν είσαι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν έχεις ε, το καθεστώς του συνεδεμένου κράτους, περιορίζεσαι μόνο στον ορίζοντα 2020 και οποτεδήποτε ας πούμε, το, η συζήτηση βγαίνει από τον ορίζοντα 2020 πρέπει να διαπραγματευτείς χωριστά. Καλή περίπτωση λοιπόν το παράδειγμα του διαστήματος ε, για το πόσο περιπλέκεται η ζωή σου αυτή τη στιγμή δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τη σύνδεξη, ο Γκέορκ την ανέφερε, την κοιτάξαμε ήδη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τμήμα ΙΤΕΡ, αλλά και άλλες χώρες επίσης. Είναι μια διακυβερνητική συνεργασία. Ε, υπάρχουν διαφορετικές διευθετήσεις και με διαφορετικές διευθετήσεις το Ηνωμένο μπορεί να συνεργάζεται στον τομέα της σύνδεξης. Αλλά κάθε φορά θα πρέπει να υπάρχουν ε, χωριστές συμφωνίες. Και εδώ, ας πούμε, αυξάνεται ο βαθμός ε, ε, προβλημάτων, περιπλοκότητα σε σχέση με το να είσαι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σχολιάσω και κάτι άλλο. Το θέμα που αναφέρατε είναι πολύ σημαντικό. Και για το Ηνωμένο Βασίλειο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θα κερδίσουμε και θα χάσουμε από τον Brexit. Για την έρευνα είναι η πιο ξεκάθαρη περίπτωση αμοιβαίου κέρδους. Ε, δεν είναι μόνο το θέμα του προϋπολογισμού, γιατί εδώ δεν υπάρχει κέρδος ή ζημία. Αλλά έχει σημασία η ερευνητική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσο πιο μεγάλος είναι ο χώρος που καλύπτει η ερευνητική περιοχή, τόσο περισσότερες, περισσότερα ωφέλη έχουμε, ε, γιατί η έρευνα γιατι η ερευνα συντελει στην ανάπτυξη. Αν φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ηνωμένο Βασίλ, θα κοστίσει αυτό, θα είναι επιζήμιο αυτό και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί θα έχουμε ένα μικρότερο χώρο έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με λιγότερη κινητικότητα, με λιγότερη αριστεία, με περισσότερους περιορισμού. περιορισμούς. Η έρευνα είναι, σαφ, είναι σαφώς ένας τομέας όπου θα μπορούσαμε να προσπαθήσουμε ότι έχει νόημα και για τους δύο το να βρουν μία διευθέτηση που θα προσωμιάζει τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, για τα νούμερα. Για αυτά που είπαμε, γιατί δεν τα δώσαμε πριν το δημοψήφισμα. Τα είχαμε τα νούμερα αυτά. Αλλά δεν είναι εύκολο να πείσεις με αναλυτικές μελέτες. Φυσικά δεν είναι δικαιολογία. Υπήρχαν αυτές οι μελέτες πάντως. Θα πρέπει να έχουμε μια νέα συμφωνία. Προφανώς. Θα πρέπει να αφήσουμε πίσω μας το παρελθόν και να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση για το μέλλον. Στον τομέα της έρευνας υπάρχει χώρος για μια ειδική σχέση που θα μας εξασφαλίσει αμοιβαία κέρδη. Ελπίζω να μην το χρησιμοποιήσουν αυτό το επιχείρημα όλοι ως διαπραγματευτικό χαρτί. Επεκταθώ λίγο περισσότερο σε ένα σημείο που έθιξε συνάδελφος, πρωτού δώσω πάλι το λόγο στον Γκέορκα. Όταν αναφέρθηκε στην περίπτωση της Ελβετίας, Ξέρετε ότι η Ελβετία το 2014 διεξήγαγε ένα δημοψήφισμα όσον αφορά τις ποσοστώσεις στην ελευθερία κυκλοφορίας. Σταμάτησε όμως τότε η συζήτηση στον τομέα της ενέργειας και δεν είναι ότι αποκλείστηκαν από τον ορίζοντα 2020, αλλά σχεδόν υποβαθμίστηκε το καθεστώς τους και μειώθηκαν πάρα πολλοί αιτήσει από την Ελβετία, μια χώρα η οποία διεξάγει πολύ σημαντική έρευνα και ήταν ουσιαστικά ένας από τους παράγοντες που τους έκανε να ξανασκεφτούν λίγο τη στάση τους, επειδή μειώθηκε τόσο δραστικά και απότομα η χρηματοδότησή τους από την Ευρώπη όσον αφορά ερευνητικά προγράμματα. Ελπίζω ότι και άλλες κυβερνήσεις βλέποντας το παράδειγμα αυτό, ενδεχομένως να συνετιστούν κάποια στιγμή, ενδεχομένως να τους απασχολήσει λίγο αυτό, να δώσω τώρα το λόγο στον συνάδελφό μου. Σας παραπέμπω σε μια έκθεση που δημοσιεύτηκε αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με την Επιτροπή σας, όπου αναφερόμαστε ξεκάθαρα στον τομέα της ενέργειας. 130 σελίδες απαριθμεί η έκθεση αυτή. Προφανώς δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες. Τα βασικά πορίσματα όμως της μελέντης, όπως και για άλλους τομείς, είναι ότι οι επιπτώσεις στην ε, Ευρώπη των 27 πλέον ε, από την ε, αποχώρηση του Μένου Βασιλείου στον τομέα της ενέργειας θα είναι συγκεκριμένες και περιορισμένες. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την περίπτωση της Ιρλανδίας, Οι σχέση της με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις υπόλοιπες 26 δηλαδή. Το ζήτημα αυτό θα είναι αρκετά ευαίσθητο και θα μας επιτρέψει ενδεχομένως να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένε εξειδικευμένε συμφωνίε μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένου Βασιλείου, σε άλλου τομεί όπω η Ευρατόμ ή η συμμετοχη στην αγορά. Τα βασικά ωφέλη, αν θέλετε, που θα μπορούσαν να προκύψουν για το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ότι μπορεί να αποτελέσει ένα ξεχωριστό εταίρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως για την Ευρατόμ θεωρούμε ότι θα είναι πολύ πολύπλοκες ε, οι διαπραγματεύσεις, ιδίως όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία της Ευρατόμα. Πρέπει ε, να δούμε επίσης ποιες συζητήσεις θα πρέπει να γίνουν στον Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη σχέση που θα έχει με την Ευρατώμα στο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ. Να προσθέσω κάτι όχι ως προεδρεύων της σημερινής συνεδρίασης, ε, ως απλό μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όλοι εμείς που λυπούμεθα για το Brexit, ουσιαστικά βλέπουμε μία δυνατότητα για να ανατραπεί η κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσφέρει μία νέα συμφωνία, μία άλλη συμφωνία στο Μένο Βασίλειο. Αυτή είναι η μόνη εναλλακτική που έχουμε, η μόνη δυνατότητα για να ανατρέψουμε τα κακό κείμενα. Και είναι πολύ σημαντικό για μας να αναγνωρίσουμε την κατάσταση και να μιλάμε περισσότερο για τις αρνητικές συνέπειες που το Brexit θα έχει στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το να μιλάμε συνεχώς για τα αρνητικά που θα επιβαρύνουν το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτό δεν εξυπηρετεί πάρα πολύ τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως, η σημερινή συζήτηση μας έδωσε πολλές χρήσιμες πληροφορίες. Πάντως, η δική μου πρόταση μάλλον δεν είναι πολύ εύκολο να ευοδοθεί. Πάντως δεν εγκαταλείπω την ελπίδα. Είμαι Γερμανός. Χάσαμε τη μάχη της Βρετανίας, ευτυχώς θα έλεγα. Νομίζω ότι θα πρέπει να κερδίσουμε τώρα τη μάχη για την Βρετανία. Κυρίε και κύριοι, αυτό ήταν το τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Υπάρχει κάτι το οποίο θέλετε να γύρετε στα πλαίσια των διαφόρων. Όχι. Ολοκληρώνεται λοιπόν τη σημερινή συνεδρία. Σας ευχαριστώ.